συνεδρίαση. Πάρα πολύ ωραία. Το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξή μας είναι η ανταλλαγή απόψεων με την Ουγγρική Προεδρία στο τομέα των μεταφορών. Και θα ήθελα να σας παρουσιάσω τον ε, Υφυπουργό ε, Μεταφορών, τον κύριο Πάουλ Βόρνερ. Είχα την ε, τιμή να τον συναντήσω ανεπίσημα πριν ε, από την έναρξη της ε, Ουγγρικής Προεδρίας. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην Επιτροπή Τουρισμού και Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προσβλέπουμε στη συνεργασία μας το επόμενο εξάμηνο. και θα θέλαμε να ακούσουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα όσα θα μας πείτε σήμερα το απόγευμα για το πρόγραμμα της Ουγγρικής Προεδρίας. Κανονικά έχετε εσείς το λόγο, μιλάτε και μετά δίνουμε το λόγο στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων, συντονιστές και ακούμε και όλα τα μέλη τα οποία έχουν να κάνουν κάποια ερώτηση. Σας καλωσορίζουμε για άλλη μια φορά και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή για μένα που μπορώ να εκπροσωπήσω τη χώρα μου εδώ ενώπιόν σας και ε, θα σας παρουσιάσω το πρόγραμμα της Προεδρίας και τις προτεραιότητές μας. Είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι η Ευρώπη θα κρατήσει τη θέση της στην παγκόσμια, στην σκηνή ε, μονάχα εάν μπορέσει να ανταπεξέλθει στις ε, τεχνολογικές εξελίξεις και ε, εάν και εφόσον δώσει νέες απαντήσεις στον τομέα των μεταφορών. Πρέπει να είμαστε ισχυροί και ανταγωνιστικοί. Οι μεταφορές είναι ένας βασικός τομέας για τις οικονομικές εξελίξεις οι μεταφορές χερσαίες, αέριες, θαλάσσιες αποτελούν ε, την κινητήρια δύναμη της οικονομίας μας, του πλούτου μας. Πέραν όμως τις οποιοδήποτε οικονομικές πτυχές υπάρχουν ε, στόχοι βιωσιμότητας ε, και προστασίας του περιβάλλοντος. Η Ουγγρική, η Ουγγρική Προεδρία συγχαίρει τις προηγούμενες ε, προεδρίες και είναι ιδιαίτερα ευγνώμων προς προεδρίες αυτές γιατί ε, εφάρμοσαν ε, τα προγράμματα και εμείς, τα οποία εμείς θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε. Για να υλοποιήσουμε τους στόχους μας πρέπει να πω ότι θα στηριχθούμε στη στενή συνεργασία όλων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να πω με λίγα λόγια το πρόγραμμα της Ουγγρικής Προεδρίας. Ας ξεκινήσουμε με τις χερσαίες μεταφορές. Ξέρετε ότι η οδηγία για την Ευρωβινιέτα εγκρίθηκε με πολύ μικρή πλειοψηφία στο Συμβούλιο. Αυτό το γεγονός ε, αφήνει πολύ ελάχιστα περιθώρια ελιγμών στην Προεδρία για, να, για τον τρόπο με τον οποίο θα συζητήσουμε τα θέματα αυτά στο, με το Κοινοβούλιο. Εάν ένα κράτος μέλος αλλάξει την, ε, τις απόψεις του στο Συμβούλιο, θα δημιουργηθεί μια μειοψηφία που θα μπλοκάρει τις όλες διαδικασίες. Ξεκινήσαμε από τη Βελγική Προεδρία και τώρα η δική μας ε, ε, Προεδρία, σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα ήθελε να ολοκληρώσει τις ε, διαπραγματεύσεις σε αυτό το τόσο ευαίσθητο τομέα. Μέχρι στιγμής έχουμε καταλήξει σε μία συμφωνία, σε κάποιες συμβιβαστικέ ε, προτάσεις που ελπίζουμε ότι θα ε, επιτευχθεί συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσα στα πλαίσια της ε, δεύτερης ανάγνωσης. Επίσης για τις χερσαίες, ελπίζουμε ότι θα κλείσει αυτός ο φάκελο με τις χερσαίες με τη μεταφορές. Οι, οι αποφάσεις του Συμβουλίου Υπουργών Μεταφορών της Δευτέρας Δεκεμβρίου επέτρεψαν ε, στην Ουγγρική Προεδρία να προχωρήσει σε δεύτερη ανάγνωση και να, ε, να ευελπιστούμε ότι θα κλείσουμε το θέμα αυτό μέχρι το καλοκαίρι. Επίσης, θέλουμε να καταλήξουμε σε μια συμβαστική λύση ανάμεσα στα τρία κοινοτικά όργανα. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να αναδιατυπώσουμε το πρώτο σιδηροδρομικό πακέτο. Υπάρχει στις 16, στη συνάντηση του Συμβουλίου στις 16 Ιουνίου διατυπώθηκε μια γενική προσέγγιση και θέλουμε να ε, περιορίσουμε τις ε, διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Αυτό θα γίνει, θα γίνει στις 16 Ιουνίου και η επόμενη Προεδρία πιστεύουμε ότι θα ολοκληρώσει το έργο. Επίσης ε, η, η εσωτερική ναυσιπλοεία, το πρόγραμμα ΝΑΙΑΝΤΕΣ, ε, για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ελπίζουμε ότι εάν ε, λάβουμε σοβαρά υπόψη μας τα θέματα εσωτερικής ναυσιπλοείας, αν τα προωθήσουμε, ε, θα έχουμε σημαντικό πλεονέκτημα, διότι πρόκειται για μία βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον ε, μέθοδο μεταφοράς. ...6 με 8 ε, Απριλίου 2011 στο Έστεργουμ θα οργανώσουμε μία συνάντηση ε, των Υπουργών ε, στο ε, που θα ασχοληθεί με τα θέματα εσωτερικής ναυσιπλοείας. Κυρίως θέματα χρηματοδότησης ε, και προώθησης των, της χρησιμοποίησης των εσωτερικών υδάτων. όλα αυτά θα προωθηθούν μέσω του προγράμματος ΝΑΙΑΔΕΣ, Το 2011, την Άνοιξη πιο συγκεκριμένα, το Κοινοβούλιο θα... Η θα ε, δημοσιοποιήσει την, ε, μια έκθεση προόδου για το Ναϊάδες και ελπίζουμε ότι τον Ιούνιο του 2011 στο Συμβούλιο των Υπουργών θα υιοθετηθεί και ε, το τροποποιημένο πρόγραμμα Ναϊάδες. η αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών και αναθεώρηση των σχετικών οδηγιών έχουν ε, δρομολογηθεί για το Μάρτιο του 2011 και θα γίνει και μια ανακοίνωση της Κομισιόν. Αυτά είναι θέματα τα οποία θα θέλαμε να συμπεριληφθούν στη μερίσια διάταξη των τεχνικών συναντήσεων, έτσι ώστε να ληφθεί μια απόφαση επίσημη πλέον στο Συμβούλιο Υπουργών στις 16 Ιουνίου. Ε, οι εσωτερικές μεταφο θαλάσσιες μεταφορές για μας είναι πάρα πολύ σημαντικές, όπως επίσης και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Και όλα αυτά ε, καλύπτονται από την περιφερειακή πολιτική του Δούναβη. Έχουν γίνει μελέτες σκοπιμο, ε, ε σκοπιμότητας, οι οποίες ολοκληρωθούν και το 2011 και μετά θα προχωρήσουμε και στην υλοποίηση των διαφόρων έργων υποδομής. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Δούναβης αποτελεί ένα ιδιαίτερα περίπλοκο περιβαλλοντικό, περιβαλλοντικά σύστημα. Γι' αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ιδιαίτερα σφαιρικά και ολοκληρωμένα μία βιώσιμη περιοχή για τον, στο Δούναβι θα αποτελέσει ένα στοιχείο κλειδί για την συνεργασία ανάμεσα στις, ε, στις χώρες της περιοχής και για να συντονίσουμε τις μεταφορές θα πρέπει να έχουμε ε, διαλειτουργικά συστήματα επικοινωνίας, ε, θα, έχουμε, θα πρέπει να έχουμε συστήματα ε, συντονισμού και ελέγχου των μεταφορών, τα οποία να είναι εναρμονισμένα σε όλη την περιοχή. Τώρα, όσον αφορά τα οριζόντια θέματα, θα θέλαμε να ασχοληθούμε με δύο θέματα στρατηγικής σημασίας, πολύ σημαντικός φάκελος για μας. 2010-2012 λευκή βίβλος για την πολιτική μεταφορών. Πιστεύουμε ότι ο τομέας μεταφορών είναι καθοριστική σημασίας για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει άμεσες, άμεση συνέπειες στην ανταγωνιστικότητα της περιοχής, εξασφαλίζει κοινωνική και οικονομική συνοχή και ε, ενισχύεται και η ενιαία αγορά. Επομένως, στην επόμενη δεκαετία και τα επόμενα χρόνια γενικότερα, θα θέλαμε να ε, υλοποιήσουμε μια πολιτική μεταφορών που να λαμβάνει υπόψη τις διαφορές που υπάρχουν, αλλά και την ε, κοινωνική, και την κοινωνική συνοχή, η οποία θα αμβλύνει τις διαφορές αυτές. Η ανακοίνωση της Κομισιόν θα δημοσιευθεί τον Μάρτιο του 2011. Υπήρχε μια αναβολή, υπήρξε μια αναβολή ε, γιατί η Κομισιόν ε, ήθελε να το να συνδυάσει αυτό με την ε, ανακοίνωση που αφορά την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα στην Ευρώπη. και αυτά όλα θα ε, συζητηθούν στο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών της 16ης Ιουνίου. Τώρα, όσον αφορά την ε, αναθεώρηση των ten ε, του προγράμματος TEN-T, πιστεύουμε ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στις υπόλοιπες, στην υλοποίηση των γενικότερων στόχων μας, εάν δεν ολοκληρώσουμε την αναθεώρηση του προγράμματος για τα TEN-T. Είναι πεποίθησή μας επομένως ότι όταν ε, σχεδιάζουμε την μελλοντική ε, φάση του προγράμματος TEN-T θα καλύψουμε τα κενά και θα πετύχουμε μια γεωγραφική ισορροπία. Σαν βασική αρχή θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η Κομισιό να ζητήσει τη συνεισφορά και τη συμμετοχή των ε, κρατών μελών στην αναθεώρηση του προγράμματος TEN-T και στην λήψη των σχετικών αποφάσεων η ανεπίσημη συνάντηση των Υπουργών Μεταφορών στις 7 και 8 Φεβρουαρίου θα ασχοληθεί με αυτά τα διευρωπαϊκά δίκτυα και πιο συγκεκριμένα με τη μεθοδολογία και την χρηματοδότηση του προγραμματισμού των δικτύων αυτών. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχουμε κατά νου, οι προτάσεις θα δημοσιοποιηθούν δημοσιευθούν για το TNT, θα δημοσιευθούν ε, από την Κομισιόν τον Ιούλιο. Επομένων, επομένως, μάλλον οι Πολωνοί θα διαπραγματευθούν ε, τα διάφορα θέματα αυτά. Τώρα, στις αεροπορικές μεταφορές ε, δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα για την ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού ουρανού. Χρειάζονται πολλά πράγματα για να, για να ολοκληρωθεί ε, αυτή η δημιουργία των ευρωπαϊκών εθέρων. Πρέπει να συμπληρώσουμε το SES, e ε, τα, θα πρέπει να ολοκληρωθεί ο, ο αποτελεσματικός να ολοκληρωθεί, να ολοκληρωθεί ένας αποτελεσματικός τρόπος διαχείρισης των, των ε, εναερίων μεταφορών. Θα Ζητηθεί στις 3 και 4 Μαρτίου στην Βουδαπέστη. Και θα εστιάσουμε την προσοχή μας στην διαχείριση των νέων αεροπορικών διαδρόμων και την εφαρμογή του SES 1 e και 2 όπως επίσης ε, και το πώς ε, οργανώνουμε ένα λειτουργικό εθέρα και ε, πόσο, οργανώ, πως θα λάβουμε υπόψη μας τα επόμενα πώς συνδυάζεται ο Σίζαρα το σίζαρα με τα επόμενα συστήματα. Στην παρούσα φάση του Ενίου ευρωπαϊκού ουρανού πρέπει να προετοιμαστούμε για την φάση ανάπτυξης του προγράμματος ΣΥΖΕΡ και είναι σημαντικό το νέο σύστημα διαχείρισης ενέργειας κυκλοφορίας να γίνει ανταγωνιστικό. Αναμένουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αρχές πολιτικής αεροπορίας των ΗΠΑ να αρχίσουν σε θέματα ανάπτυξης και έρευνας πρόγραμμα συνεργασίας στην Άνοιξη. Επίσης, αποδίδουμε μεγάλη σημασία στο θέμα των καλών σχέσεων όσον αφορά σε επίπεδο διεθνές την πολιτική αεροπορία. Θα υπογράψουμε μία, μάλλον θα εγκρίνουμε μία απόφαση του Συμβουλίου για συνεργασία μεταξύ ημών και ΙΚΑΟ. Σε θέματα συνεργασίας με τρίτες χώρες θα προχωρήσουμε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τις προτάσεις Επιτροπής. Η Ουγγρική Προεδρία μόλις υποβάλλει στην πρόταση η Κομισιό θα προβλέψει την ε, εντολή για την ε, ε, συμφωνία συνεργασίας την Μόλοβα, καθώς και μία συμφωνία καμποτάζ με την Ελβετία. Αναμένουμε επίσης προτάσεις Επιτροπής για την προσχώρηση της Ισλανδίας και της Νορβηγίας στον Ευρωπαϊκό Εναέριο Χώρο. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να εγκρίνουμε στο τομέα αυτό και απόφαση του Συμβουλίου και υπάρχει και πρόοδος για μια συμφωνία συνεργασίας και με την όπως ξέρετε, σε θέματα Επίσης, ε, τελωνιακά θα έχουμε συνεργασία, δεδομένου ότι εμείς είμαστε μια χώρα που σχεδόν περιβάλλεται ε, από πολλές άλλες χώρες. Έχουμε και την εμπειρία της Βελγικής Προεδρίας, των Βέλγων ε, συναδέλφων που θα μας βοηθήσουν και διάρκεια της Προεδρίας μας και βεβαίως εμείς θα ακολουθήσουμε τις εργασίες της Βελγικής Προεδρίας για την αναθεώρηση της, ε, του κανονισμού που αφορά την Διεθνή Οργάνωση Ασφαλείας των Θαλασσίων Μεταφορών. Και ελπίζουμε να καταλήξουμε και σε άλλη συμφωνία τον Μάρτιο. Τώρα, όσον αφορά τον τομέα των ε, εξοπλισμών, στον τομέα της ναυσιπλοείας. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Θέλουμε ή να έχουμε μία, προωθήσουμε σε μία γενικότερη προσέγγιση, ακόμη και να καταλήξουμε συμφωνία Συμβουλίου στο Συμβούλιο του μηνός Ιουνίου. Επίσης, θα θέλαμε να επιτύχουμε και άλλες συμφωνίες στα πλαίσια των μεταφορών μετά από την πρώτη ανάγνωση του Συμβουλίου. Κυρίες και κύριοι, ξενορίζω πάρα πολύ καλά ότι μεταξύ των κρατών μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής θα πρέπει να έχουμε καλή συνεργασία για να επιτύχουμε στις στόχους μας και τη διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας. Πρέπει να σας πω ότι εμείς είμαστε ανοιχτοί για συνεργασία, για διαβούλευση και για λογικές συμφωνίες. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Περιμένω τις ερωτήσεις και είμαι σίγουρος ότι η συνεργασία μας κατά τη διάρκεια του παρόντος εξαμήνου θα είναι επικοδομητική. Σας ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ Βόλνερ. Πρώτα απ' όλα, ερωτήσεις εκ μέρους των συντονισμών. Θα ήθελα να μου πείτε παρακαλώ, θα σας πω ποιοι είναι οι συνάδελφοι οι οποίοι θέλουν να λάβουν το λόγο και μετά θα ήθελα να δω ποιο άλλο θα το λόγο για να κάνω τις μαθηματικές μου πράξεις, ανάλογα με το χρόνο να δω πόσους έχουμε. Mrs. Meissner, Mrs. Lichtenberger, I don't know whether Mr. Kolicek wants... κύριος Κόλιτσεκ και ο κύριος Κόλιτσεκ θέλει. Τον προσθέτω στον κατάλληλο. And then I have Mr. Kolza, Mr. Liberatsky, Mrs. Gourmay, Mrs. Foster, Mrs. Mr. Kantian. Is there anybody else? Θέλει κανένας άλλος συνάδελφος το λόγο, ο κύριος Ουρζιάς. Anybody else? Okay. Έμεινε κανείς εκτός. Λοιπόν, αυτό είναι ο κατάλληλος των συναδέλφων. Για να έχουμε αρκετό χρόνο και να οργανωθούμε. Οι συντονιστές πρώτα, οι απαντήσεις. Οι συντονιστές έχουν τέσσερα λεπτά ο καθένας. Τέσσερα λεπτά. Με τον κύριο Γκρός θα αρχίσουμε για τέσσερα λεπτά. Κύριε Γκρός, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στο εξάμεινό σας. Οι μεταφορές όπως ξέρετε είναι ένα από τα σοβαρότερα θέματα και στο κοινοβουλίο μας και Πρόκειται για ένα θέμα κιόλα που σχετίζεται πολύ με τις προσδοκίες των πολιτών των οποίων επηρεάζεται η καθημερινή ζωή. Έχετε... Ε, υπάρχουν δύο θέματα, από τη μια η Ευρωβινιέτα και από την άλλη ο Σιδηρόδρομος που Ελπίζουμε τα θέματα αυτά να τα λύσει η Ουγγρική Προεδρία γιατί πιστεύουμε ότι αυτό θα είναι καλό για την Ευρώπη. Η Ευρωβουνιέτα δεν θα πρέπει να γίνει ένα θέμα στο οποίο να πεισμώσει το Συμβούλιο και να μην κάνει τίποτε τον να να μην κάνουν τίποτα άλλο τα κράτη-μέλη παρά μόνο να παίρνουν ε, χρήματα από τις τσέπες των πολιτών ε, τα πράγματα δεν προχωρούν όταν όμως υπάρχουν τέτοιου είδους καλές πρωτοβουλίες που βοηθούν και τα κράτη και τους πολίτες και δημιουργούν ίσως νέες ε, πηγές στο χώρο των μεταφορών και στο ε, αυξάνουν την κινητικότητα στην Ευρώπη τότε αυτό είναι καλό και το Ευρωκοινοβούλιο θα σας βοηθήσει ε, με κάθε όπως μπορεί για να προωθηθούν τέτοιου είδους ε, ε πρωτοβουλίες και το και για το σιδηρόδρομο ε, η, τα πράγματα είναι παρόμοια. Τα κράτη-μέλη δρούν σε σχέση με τους σιδηροδρόμους και ε, σαν να ήταν ο σιδηρόδρομος το κατεξοχήν εθνικό προϊόν. Ε, πράγμα το οποίο δεν βοηθάει κανέναν. Γι' αυτό λέμε ότι στο μέλλον θέλουμε ε, μια ε, ισχυρή ανοιχτή αγο... σιδηροδρομική αγορά στην Ευρώπη και αυτό θα βοηθήσει και τα κράτη και τα... τους πολίτες. Αυτά τα δυο λοιπόν Ευρωβινιέτα και σιδηρόδρομο θα πρέπει να τα προωθήσετε και ελπίζουμε να τα κλείσετε. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα θέματα. Ο νέος ευρωπαϊκός ουρανός, να ένα άλλο παράδειγμα για το πώς θα μπορούσαμε να δώσουμε κάποια σινιάλα για την, το μέλλον της Ευρώπης. Η εσωτερική ναυσιπλοεία είναι ένα άλλο πράγμα που θα μπορούσαμε να προωθήσουμε αλλά ειδικά για τους εθέρες της Ευρώπης ιδιαίτερα μετά την έκρηξη του ηφαιστείου στην Ισλανδία είδαμε πόσο δύσκολο Κόλλα και κακά είναι τα πράγματα. Γι' αυτό πρέπει να φροντίσουμε να φτιάξουμε μια Ευρώπη, τον, μια έναν ουρανό πάνω από την Ευρώπη που να μην έχει 27 συνιστώσεις αλλά που να είναι ενιαίος και αυτό το περιμένει ο πολίτης και το προσδοκά δεν θα ήθελα να συνεχίσω παρόλο που θα μπορούσα να αναφέρω και άλλα θέματα κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ θα κλείσω γιατί τελειώνει ο χρόνος μου εύχομαι καλή επιτυχία Πρόεδρος ξεπεράσατε το χρόνο σας κατά δύο δευτερόλεπτα λέει ο Πρόεδρος κάνει να τα καταφέρουν κι άλλοι τόσο καλά Παρακαλώ En uh, veel succes, zou ik zeggen. U uh, hebt een uh, belangrijke uitdaging voor de boeg. Het er zijn belangrijke dossiers die op de agenda staan. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ε, κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε. Πραγματικά αναφέρατε πολλών, πολλά πολύ σημαντικά θέματα. Ε, εκ των οποίων θα ήθελα να αναφέρω δύο. Ε, θέματα τα οποία για μένα έχουν τη μεγαλύτερη σημασία. Η Ευρωβινιέτα είναι το ένα και οι διασυνοριακές παραβάσεις είναι το άλλο. Νομίζω ότι τα θέματα Αυτά ε, πράγματι είναι θέματα που α, εντάσσονται στην καθημερινότητα του πολίτη και που περιμένει ο πολίτης να επιληθούν. Ξέρω γιατί είμαι εισηγητής για την Ευρωβινέτα ότι τα πράγματα στο Συμβούλιο είναι πάρα πολύ δύσκολα για το θέμα αυτό. Θα, εμείς θα επιμείνουμε, θα προσπαθήσουμε να πιέσουμε το Συμβούλιο να προχωρήσει ε, με, την Ευρω... με την οδηγία αυτή για την Ευρωβινέτα. Θα επιμείνουμε για τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων. Θα επιμείνουμε για κάποιες ε, πρωτοβουλίες πρέπει να αναλυφθούν τα επόμενα χρόνια για την ε, εσωτερικοποίηση αν θέλετε των εξωτερικών του εξωτερικού κόστους θα επιμείνουμε για όλα αυτά Βεβαίως υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία σχετίζονται με το απότερο αν θέλετε μέλλον. Μιλήστε για τον σιδηρόδρομο, για τη χρηματοδότηση των μεταφορών στην Ευρώπη, για το πρόγραμμα TNT και τις κατευθυντήριες γραμμές του και το νέο ε, δημοσιονομικό πλαίσιο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Α, πράγματι εύχομαι καλή επιτυχία για όλα τα θέματα αυτά, αλλά θα ήθελα να παρακαλέσω να λάβετε υπόψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε όλα αυτά, το οποίο θα ήθελε αν είναι δυνατόν να εμπλέκεται ε, ήδη εξ αρχής στη συζήτηση αυτών των θεμάτων. Γιατί τελικά υπάρχουν Έχουμε κι εμείς ένα ευρωπαϊκό όραμα. Έχουμε ένα όραμα για το μέλλον της Ευρώπης, το μέλλον των μεταφορών στην Ευρώπη που είναι πέρα από τα εθνικά σύνορα και γι' αυτό θα αγωνιστούμε. Θέλουμε να υπάρχουν ε, να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο στην Ευρώπη για τις μεταφορές το ίδιο και όχι μόνο στη Χέρσον θέλετε αλλά και στη θάλασσα και στον αέρα ο ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός που αναφέρατε νομίζουμε ότι ε, σε αυτά θα μπορούσαμε πάρα πολύ καλά να συνεργαστούμε το Συμβουλίο και εμείς εκ μέρους των φιλελευθέρων η κυρία Μάισνερ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ και χαίρομαι που βρίσκεστε εδώ στο Κοινοβούλιο. Αναφέρθηκαν πολλά πράγματα, εγώ θα περιοριστώ σε τρία. Στην Ευρωβινιέτα που ανέφερα η Ευρωβινιέτα είναι ένα θέμα βέβαια, αλλά εγώ θα ήθελα να αναφέρω άλλα τρία. Πρώτα-πρώτα τις θαλάσσιες μεταφορές και τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές. Ιδιαίτερα για την εσωτερική ναυσιπλοεία, θα ήθελα να δω τι έχετε κατά νου. Μιλήστε για τις υποδομές, για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Αν αναφερθήκατε στην περιοχή του Δούναβη, Ξέρετε πολύ καλά ότι η στρατηγική του Δουνάβη, του Δουνάβη αυτή τη στιγμή ε, απασχολεί το Κοινοβούλιο. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι πρωτός παντού ο Δούναβης. Αλλά θα... Γι' αυτό ρωτάω τι φαντάζεστε, γιατί θα πρέπει να δείτε και το κατά πόσον κάποιος ο αποταμός είναι πλωτός, που υπάρχουν όρια, που υπάρχουν ευκαιρίες για το μέλλον. Δε... Είπατε επίση ότι δεν υπάρχουν, δεν έχετε ε, θαλάσσιες μεταφορές εσείς σαν χώρα, σαν Ουγγαρία. Ε, ωραία, αλλά περιμένω η Προεδρία σας κάτι να κάνει και για τις ακτές ή τουλάχιστον να συζητήσει. Ε, εκείνο που είναι σημαντικό όμως για μένα είναι να, δει, να μου εξηγήσετε πώς θα αναπτύξετε οικονομικά τον Δούναβη. Μετά αναφερθήκατε στο τεντή. Είναι πολύ σημαντικό και βεβαίως <clears throat> οι άξονες μεταφορών ουσιαστικά είναι οι αρτηρίες οι υπομοδοτούν ουσιαστικά την Ευρώπη. Λοιπόν, εδώ παίζουν μεγάλο ρόλο όμως όχι μόνο οι οδικές αρτηρίες αλλά και οι σιδηροδρομικές αρτηρίες. Θα με ενδιέφερε ιδιαίτερα να μου πείτε ε, στα δίκτυα αυτά και στο ε, σιδηροδρομικό δίκτυο δίκτυο τι ε, προτίθεστε να κάνετε. Ε, θα ξέρετε ότι στην ε, Σαραγκόσα ε, επί Ισπανικής Προεδρίας είχαν γίνει σχετικές συζητήσεις και το επόμενο θέμα που θα ήθελα να θίξω είναι κάτι που δεν το αναφέρατε καθόλου που όμως νομίζω ότι συζητήθηκε από όλου. είναι η αεροπορική ασφάλεια η ασφάλεια στις εναέριες μεταφορές αλλά και στα αεροδρόμια. Είμαι σκιώδη συγγήτρια για συναφή θέματα και ξέρετε πολύ καλά ότι τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες απόπειρες τρομοκρατικών ενεργειών βλέπουμε στα διάφορα αεροδρόμια. Θα ήθελα να ξέρω τη θέση της Ουγγρικής Προεδρίας για τα, το θέμα αυτό. Αυτά είναι τα τρία θέματα λοιπόν που Αυτά ήθελα να θέσω εγώ. Κατά τα άλλα εύχομαι καλή συνεργασία. Η κυρία Λίχτερμπεργκερ τώρα εκ μέρους των Πρασίνων για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ τον Υπουργό για την παρουσία του προγράμματος της Προεδρίας. μεγάλο και φιλόδοξο το πρόγραμμα. Είναι πολύ καλό να δούμε τέλος πάντων τι θα επιτευχθεί από όλα αυτά. Τέλο πάντων, για τον Δούναβη τώρα, όπως ανέφερε και η συνάδελφος, θα ήθελα και εγώ να ζητήσω να μας πείτε μερικά παραπάνω πράγματα. Πώς φαντάζεστε αυτή τη στρατηγική του Δούναβη, πώς θα βελτιώσετε την αναψυπλοεία στο Δούναβη. Είναι ιδιαίτερα πεπαλαιωμένη υποδομή η ΑΚΙ και ε, υπάρχουν διακοπές στις συνδέσεις αν θέλετε και καταλαβαίνετε ότι ε, πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχουν συνδέσεις και για τις εμπορευματικές μεταφορές προφανώς. είμαστε υπέρ του να κάνουμε προσπάθειες να προσαρμοστούν τα σκάφη προς τον ποταμό και να μην περιμένουμε ε, να προσαρμοστεί ο ποταμός στα σκάφη ε, θέλω να μας πείτε μερικά πράγματα για αυτό τα river adapted ships Γι' αυτό το μοντέλο επίσης κάτι τι άλλο θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα στις θαλάσσιες μεταφορές. Ξέρω ότι δεν έχετε ε, θάλασσα, αλλά πολλές φορές αυτοί οι οποίοι δεν είναι ε, μπλεγμένοι σε ορισμένα θέματα ε, να ε, είναι καλύτεροι στη διευθέτηση των θεμάτων αυτών και για την ε, και θα ήθελα αν είναι δυνατόν πέρα, να, να φροντίσει η ε, Ουγγρική Προεδρία να υπογραφεί το πρωτόκολλο με τις Άλπεις για το σιδηρόδρομο τώρα στην Επιτροπή Μεταφορών για το τριμερές για το τρίγωνο των τριών χωρών είχαμε συζητήσει και ένα είδο σιδηροδρομικής σύνδεσης εκεί και τέλος το θέμα της του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού ακόμη και να έχει δημιουργηθεί αυτό το παιδάκι είναι ακόμη πάρα πολύ μωρό θα πρέπει να προωθηθεί η υπόθεση αυτή και μάλιστα γρήγορα. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Βαντάλεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να καλωσορίσω και εγώ τον Υπουργό εδώ στην Επιτροπή μας. Δεν νομίζω ότι θα εξαντλήσω και τα τέσσερα λεπτά. Ένα θέμα θέλω να θίξω εγώ. Καταρχάς όμως να σας συγχαρώ γιατί επιστήσατε την προσοχή μας στα θέματα εσωτερικής ναυσιπλοείας. Είναι πάρα πολύ σωστό, πιστεύω, να θίξουμε αυτό το θέμα και να εξετάσουμε αυτό το θέμα μεταφοράς, που είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, για όλους μας και νομίζω ότι ο τρόπος που αντιμετωπίζετε το θέμα αυτό είναι επίσης πολύ καλός. Η κυρία Μάισνερ το είπε, όταν μιλάμε για εσωτερική ναυσιπλοεία μιλάμε πολύ συχνά για υποδομές αλλά το πρόβλημα υπάρχει. Υπάρχουν κάποιες αδυναμίες, τις οποίες έχουμε συζητήσει ήδη. Και η ερώτησή μου, Πρόεδρε, είναι τι θα κάνετε για τι θα κάνετε για να βρούμε λύσεις, συγκεκριμένες πρακτικές λύσεις και ε, να δημιουργηθούν τα απαραίτητα φράγματα για να ε, υπάρχουν, να υπάρχει μια πραγματική σύνδεση, διότι μιλάμε για τα μεγάλα ποτάμια. Ε, Αλλά μην ξεχνάμε ότι είχαμε και το ατύχημα στο Ρήνο με την Το σύστημα ασφάλειας του σκάφους λειτουργήσε καλά, άρα δεν ε, θρυνήσαμε μια καταστροφή. Αλλά θα πρέπει να βρούμε λύσεις και για τα ε, ρεύματα, για, τα ρεύματα που, δηλαδή για τις... Ε, για, τα μέρη του, των, των εσωτερικών υδάτων όπου, ε, τα, τα οποία ρέουν γρήγορα. Θυμόσαστε το ατύχημα του Excelsior πριν από πέντε χρόνια και είχαμε πει ότι θα δημιουργήσουμε ένα σύστημα διάθεσης ε, των ε, ναυαγίων στο Ρήνο. Θα το συζητήσετε για αυτό το θέμα στο Άστεργκούνο. Έχετε να προτείνετε μια λύση. Τέλος μας σας εύχομαι καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ. Μόνο δύο πολύ σύντομες ερωτήσεις. Όσον αφορά τις οδικές μεταφορές, αναφέρατε κύριε Υπουργέ ότι σας ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα το ένα πρόγραμμα δικής ασφαλείας. Τι έχετε να πείτε για τα οδικά ατυχήματα που γίνονται εκτός συνόρων πολλές φορές. Επίσης, στα πλαίσια του πρώτου πακέτου σιδηροδρομικών μεταφορών, θα ενισχύσετε σε τοπικό περιφερειακό επίπεδο την διασύνδεση φερρυππιν μεταξύ Αυστρίας, Ουγγαρίας. Όταν επίσης ε, επισκεφθήκαμε το τρίγωνο Τσεχοσλοβακίας, Ουγγαρίας, Αυστρίας είδαμε τι σημαίνει. Τώρα, στα πλαίσια του ΣΥΖΑΡ θα αυξήσετε την ε, ασφάλεια. Τι θα κάνετε επίσης μεταξύ ε, των Επίσης, τις εσωτερικές πλωτές οδούς. Τι θα κάνετε με το θέμα του Δούνα και του Ελμ. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, εάν θέλετε μπορείτε να απαντήσετε, αν μπορείτε να απαντήσετε σε 10 λεπτά έχει καλώς σε αυτό την πρώτη σειρά ερωτήσεων και μετά θα προχωρήσουμε. Έχετε λοιπόν το λόγο αν θέλετε να απαντήσετε στο πρώτες ερωτήσεις που τέθηκαν. Σας ευχαριστώ. Η ιδέα της ε, συνέχειας ε, του follow-up μετά από αυτά τα οποία έκαναν η Ισπανική και η Βελική Προεδρία ήταν από τις πιο σημαντικές ιδέες. Άκουσα επίσης διάφορες ερωτήσεις ε, για την οδηγία που αφορά την Ευρωβινιέτα και τη δυνατότητα δεύτερης ανάγνωσης. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι σημαντικό και αν υπάρξει συμφωνία θα έχουμε ένα σύστημα πιο διαφανές. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσει να ολοκληρωθεί η δουλειά μετά από η συμφωνία μετά από χρόνια δουλειά. Πιστεύω λοιπόν ότι ακόμη και αν υπάρξει περιορισμένη σε συμφωνίας θα έχουμε κάνει κάτι το πολύ συναμαντικό. Θα δούμε πώς θα διευθετήσουμε τα πράγματα. Καλύτερα είναι να καταλήξουμε σε μια συμφωνία όπου και ο χρήστης θα πληρώνει κάτι και ο ρηπένα θα πληρώνει κάτι παρά να μην καταλήξουμε καθόλου σε συμφωνία. Και βεβαίως αν δεν είναι πάρα πολύ ε, επιτυχής η συμφωνία καταρχάς μπορούμε να την αναθεωρήσουμε και να την βελτιώσουμε βάσει της εμπειρίας σε μια δεύτερη φάση. Όσον αφορά την αναδιατύπωση του πακέτου μέτρων που αφορά τις υδροδρομικές μεταφορές, θα πρέπει να σας πω ότι στις μεταφορές τα πάντα ε, αλληλοσυνδέονται μεταξύ τους. Αν μιλούμε για την ε, Ευρωβινιέτα και για την αρχή του οριπένων πληρώνει, ίσως κατορθώσουμε να έχουμε μία ουδέτερη προσέγγιση, αν θέλετε, μεταξύ των σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. Πράγμα που σημαίνει θα προστατεύσουμε και το περιβάλλον και θα ικανοποιήσουμε και αυτούς οι οποίοι μιλούν για ηχορύπανση. Πολλά μέλη επίσης ανέφεραν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα της αναδιαπτώσης της ε, πακέτου μέτρων για τις αδικές μεταφορές, διότι διακυβεύονται πολλά ε, διασυμφέροντα πολλών κρατών. Αλλά βεβαίως θέλουμε να συναντώμεθα συχνά και ίσως ακόμη και σε εβδομαδιαία βάση για να μπορέσουμε σιγά σιγά να επιτύχουμε, επιτύχουμε συμφωνία. Και θα συζητήσουμε κάποια στιγμή και την έκθεση πρόοδου στον τομέα αυτό. <coughs> Όσον αφορά το εξωτερικό κόστος και πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια και τα έσοδα τα οποία αποκτούμε από αυτό το εξωτερικό κόστος, θα θέλαμε τα κονδύλια αυτά να χρησιμοποιηθούν από τον ίδιο τον τομέα αυτό. Πολλές φορές υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν θέλουν να επιβάλλουν μια υποχρεωτική τέτοιου είδους λύση. Προσπαθούμε σε αυτή την περίπτωση να καταλήξουμε σε συμβιβαστικές λύσεις, αλλά κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε κάποια συμφωνία να αποδεκτεί από όλου. Συμφωνώ επίσης με τον κύριο Κρός ότι όντως χρειαζόμαστε μια ισχυρή και ανοιχτή ενιαία εσωτερική αγορά και γι' αυτό είναι απαραίτητο να έχουμε την αναδιατύπωση του πακέτου για τις συνδρομικές μεταφορές. Εμείς είμαστε υπέρ μιας ισχυρής Ευρώπης και μπορεί να συνεισφέρει ο τομέας των μεταφορών πάρα πολύ. Επίση, ξετάζουμε όλα τα είδη των μεταφορών, την αυσιπλοεία, τις εσωτερικές πλωτές οδούς, την ενέργεια κυκλοφορία, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μία ισχυρή ενιαία εσωτερική αγορά με τη συνεισφορά όλων των μέσων μεταφοράς. Επίσης, οι εσωτερικές πλωτές η εσωτερική ναυσιπλοεία δεν είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να επιληθεί τμηματικά, δηλαδή δεν μπορούμε να βρούμε μία λύση μόνο για ένα ποτάμι στην Ευρώπη. Θα πρέπει να έχουμε μία λύση ενιαία για όλες τις εσωτερικές πλωτές οδούς. Επίσης θα πρέπει στα πλαίσια των ε, σχεδίων ε, ε, επενδύσεων ή την ανάπτυξη μια βιομηχανία σε μια περιοχή, να μην λάβουμε μόνο υπόψη τι συμβαίνει μόνο στην περιοχή, αλλά και να δούμε πώς θα μπορέσει να έχει κανείς πρόσβαση σε αυτή την περιοχή. Το θέμα της τάχτης ξέρουμε ότι μας απασχόλησε πέρσι πάρα πολύ και η δημιουργία των hubs είναι ένα πράγμα το οποίο επίσης μας απασχόλησε. Η Ουγγαρία και οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων θα υπογράψουν μια σχετική ε, συμφωνία που είναι σημαντική για την περιφερειακή μας ανάπτυξη. Τώρα, η οδική ασφάλεια είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις και να έχουμε πρόστιμα στην περίπτωση ε, παρανομιών, αλλά θέλουμε οι δρόμοι να είναι ασφαλείς και η οδήγηση να είναι ασφαλής. Δηλαδή, θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε αυτούς που παραβιάζουν την οδική ασφάλεια, που πίνουν και οδηγούν που τρέχουν πολύ και οδηγούν. Όλα αυτά για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την οδική ασφάλεια, επαναλαμβάνω. Η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο επίσης θα πρέπει να πάρουν μία απόφαση για το αν θα θελήσουν να συμμετέχουν επίσης στι διαπραγματεύσεις και ελπίζω ότι μέχρι τον Ιούλιο θα μπορέσουμε να πληρώσουμε τις συζητήσει για το θέμα αυτό. Τώρα, όσον αφορά τα δίκτυα TNT και τη χρηματοδότηση του τομέα των μεταφορών. Όπως ε, ξέρετε, ούτε εσείς ούτε εμείς είμαστε υπεύθυνοι για την κατάρτιση του κοινοτικού προπολογισμού. Θα θέλαμε και η Κομισιόν και το Συμβούλιο να μπορέσουν να συνεργαστούν ώστε να βρεθεί μια λύση και ο τομέας των μεταφορών να μην υποφέρει από περικοπές των κονδυλίων. Τώρα, αύξηση των κονδυλίων δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να αναμένουμε από τα κράτη-μέλη στον τομέα των μεταφορών, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα, τα διαθέσιμα κονδύλια με πιο αποδοτικό τρόπο. Ουγγρική Προεδρία πιστεύω ότι μπορεί να διαδραματίσει ρόλο βοηθώντας την Επιτροπή ώστε να της καταδεικνύουμε τις πιο σημαντικούς τα πιο σημαντικά θέματα πρέπει να συζητηθούν στον τομέα των μεταφορών, αλλά βεβαίως εάν δεν υπάρχει εκ μέρους των κρατών μελών συνένεση για ένα θέμα, όπως ξέρετε, δεν μπορούν να ληφθούν αποφάσεις. Όσον αφορά την ασφάλεια των εναερίων μεταφορών. Ο Επίτροπος Κάλλας είναι υπεύθυνο για το μεταφορές και ελπίζουμε ότι για το Συμβούλιο του Ιουνίου η Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις, αλλά και πάλι ο τομέας αυτός αποδεικνύει ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη πάρα πολλά επιμέρους θέματα για την διευκόλυνση της ε, διαχείρισης της κυροφορίας, την εξυπηρέτηση των, πελατών, των επιβατών στα αεροδρόμια, των ε, σκάνερ που υπάρχουν στα αεροδρόμια, και θα πρέπει να συζητήσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες όλα αυτά τα θέματα πριν να φτάσουμε στο Συμβούλιο και καταλήξουμε σε αποφάσει. Τα ευρωπαϊκά συμφέροντα ίσως είναι υπεράνω στον τομέα των κρατικών ε, συμφέροντων και τα δίκτυα TNT αυτό αποδεικνύουν. Σήμερα είναι πολύ σημαντικό εφόσον χρησιμοποιούμε κοινοτικά κονδύλια στον τομέα αυτό, να είμαστε προσεκτικοί και να δούμε ποια σχέδια ακριβώς μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε. Πολλές φορές βλέπουμε ότι πάντα υπάρχει ένα κενό επειδή υπάρχουν κενά, γι' αυτό υπάρχουν και φυλάξει το αυτό, γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και τα κονδύλια τα οποία χρησιμοποιούμε, να τα χρησιμοποιούμε για να καλύψουμε τα ε, κενά που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, φερρυπίν, για σημεία επαφής ε, ε, για τις διακρατικές μεταφορές. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία θα καλύψουμε ως Προεδρία μεταξύ άλλων. Όσον αφορά τον Δούναβη και την ευρύτερη περιοχή, όπως ξέρετε, έχουμε να κάνουμε με ένα πάρα πολύ ε, πολύπλοκο θέμα, δεδομένου ότι ο Δούναβης διασχίζει πολλές χώρες και από οικολογικής πλευράς θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Η διαχείριση των πλημμυρών, τα αρδευτικά έργα, επίσης είναι ενδιαφέροντα θέματα και ξεπερνούν τον τομέα των μεταφορών. Βεβαίως ότι κάνουμε και όλες οι πολιτικές μας θα πρέπει να είναι φιλικές προς το περιβάλλον ε, και θα είμαστε, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί παρά το γεγονός ότι ξέρουμε ότι η εσωτερική ναυσιπλοεία είναι πολύ πιο ήπια αν θέλετε για το περιβάλλον από τις οδικές ή άλλες μεταφορές. Θα πρέπει όμως να είμαστε προσεκτικοί, να ξέρουμε τι είδους εξοπλισμό πρέπει να έχουν τα πλοία, τι είδους καύσιμα να χρησιμοποιούν. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία εξετάζουμε και όλα αυτά θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο συμφωνίας πριν να φτάσουμε στο Συμβούλιο, δεδομένου ότι δεν μπορούμε να επιβάλλουμε τίποτα στις χώρες εάν δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ τους. Ελπίζω ότι μπόρεσα να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Έχω τώρα στον δεύτερο κατάλογό μου 7 ομιλητές. Θα αρχίσουμε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 Σαν μέλος του ΕΛΚ στην Επιτροπή, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό και την ομάδα του για, το εξαιρετικό, για την εξαιρετική παρουσίαση του προγράμματος της Προεδρίας. Ανέκαθεν ε, ρώταγα κάθε προεδρεύοντα που ερχόταν εδώ να μας πει ε, ποιες είναι οι εξελίξεις όσον αφορά τα δικαιώματα των επιβατών. Όπως έλεγα, υπήρξε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα. Λοιπόν, το θέμα των ε, δικαιωμάτων των επιβατών είναι ανέκαθεν στην ε, ημερήσια διάταξη, ήταν εδώ και πολύ καιρό στην ημερήσια διάταξη και ε, υπάρχει και μια ανακοίνωση, την οποία περιμένουμε της, από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που θα δημοσιευθεί μέχρι το τέλος του έτους και θα ήθελα να ξέρω οι προθέσεις του Συμβουλίου ποιες είναι Ελπίζουμε, μπορούμε να ελπίζουμε ότι η νομοθετική διαδικασία θα ολοκληρωθεί και οι Ευρωπαίοι επιβάτες ανεξάρτητα από τα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούν θα χαίρουν των ιδίων δικαιωμάτων. Κύριε Γκρούμερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο το σχέδιό σας και θέλουμε να δημιουργήσουμε ε, μια ισχυρότερη Ευρώπη. Ελπίζω να είδατε αυτή την δημοσίευση όλοι σας, το ε, έντυπο, το οποίο σας ε, δίνει κάποια στοιχεία σχετικά με, την, με το πρόγραμμα της Ουγγρικής Προεδρίας. Είναι πολύ ενδιαφέρον ανάγνωσμα θα έλεγα. Είτε πολύ σημαντικές οι σχέσεις, καλές σχέσεις Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Και Ήμουνα η πρώτη εισηγήτρια το 2008 για το FES όχημα, FES αυτοκίνητο και υπάρχει και ένα μνημόνιο το οποίο έπρεπε, ένα MOU το οποίο έπρεπε να είχαμε υπογράψει εδώ και καιρό Ο κύριος Σμιτ ήταν συνεισηγητής για τα θέματα των ταχυδρομικών ε, θεμάτων και δεν ξέρω, η... η Ουγγρική Προεδρία έχει την πρόθεση να επανεξετάσει το θέμα αυτό των ταχυδρομικών ε, υπηρεσιών και κυρίως ε, τις συνθήκες εργασίας των ταχυδρομικών υπαλλήλων. Μιλήσατε για τον ανθρώπινο παράγοντο, για τον ανθρώπινο πρόσωπα, κυρίως όσον αφορά τον Δούναβη. Ε, επομένως, ο Δούναβης ε, δεν είναι απλώς ε, ένα ξερό πρόγραμμα, είναι κάτι γενικότερο και παρουσιάζει μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση και στη συνάντηση αυτή στη Βουδαπέστη νομίζω ότι όλοι πρέπει να έρθουν για να δούμε τι ακριβώς εννοούμε. Ευχαριστούμε ε, για όσα είπατε και για την, ε, τα όσα έγιναν και για την στη Βουδαπέστη. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ και τον Υπουργό και θα προσπαθήσω να βγω λίγο από την Ουγγαρία. Στην ε, παρέμβασή σας επαναλάβετε τα λόγια του Βίκτορα Ρόνανα για μια δυνατή Ευρώπη. Αυτή τη δύναμη όμως μεταφορές πώς θα τη δούμε. Ποια ιδέα έχετε εσείς για να ξεπεράσετε την κρίση σε αέριες μεταφορές. Γιατί καταλαβαίνω τις δυσκολίες σας, είναι η αρχή της, ε, της θητείας σας, επομένως Τέλο πάντων ακόμα δεν ξέρετε τι θα γίνει. Για να έχουμε όμως μια δυνατή Ευρώπη πρέπει να έχουμε και μια δυνατή ιδέα. Ποια είναι η ιδέα η δυνατή αυτή που έχετε. Επίσης μιλήσατε και για διαπραγματεύσει όσον αφορά το καμποτάζ. Μπορείτε να μας πείτε λίγα πράγματα για αυτή τη διαπραγμάτευση. Αυτά και ευχαριστώ από τον προτέρων. Η κυρία Φώστερ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Υπουργό και να τον ευχαριστήσω για την τόσο πλήρη παρουσίαση του προγράμματος των επόμενων μηνών. Θα ήθελα να θίξω το θέμα καταρχάς της Λευκής Βίβλου που αναφέρεται και στο εγχειρίδιο που έχουμε στη διάθεσή μας και όσον αφορά τις αεροπορικές μεταφορές στην, στην αρχική εκδοχή της, βίβλου, της Λευκής Βίβλου είχαμε μονάχα μισή σελίδα. Επίσης αναφέρεται καθόλου το ΣΕΖΑΧ και κάπου είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και στον τομέα των αέριων μεταφορών κυρίω. Είπατε ότι θα και το όντω και καλωσορίζουμε το γεγονό ότι οργανώνεται αυτή τη συνάντηση στη Βουδαπέστη υψηλού επίπεδου το Μάρτιο και θα θίξουμε τα θέματα του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού. Ε, εμείς ε, το συζητάμε αυτό το θέμα στην Επιτροπή μας εδώ και 10 χρόνια. Και Καλωσορίζω αυτά τα οποία είπατε για την Ουγγαρία και την περιοχή σας, αλλά πραγματικά για τα FABs δεν έχουμε προχωρήσει ιδιαίτερα, κυρίως για τον αριθμό των FABs τον οποία χρειαζόμαστε γενικώ. Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση ε, και ε, ήθελα να πω κάτι για το ΣΕΖΑΡ τα ΦΑΜΣΑ συνδέονται άμεσα με τα όσα συμβαίνουν για το ΣΕΖΑ και υπάρχουν ε, πολλές ε, δημόσιες ε, επενδύσεις, πολλές μικρές επιχειρήσεις έχουν, κάνει, έχουν προχωρήσει επενδύσεις και τα πράγματα πηγαίνουν πάρα πολύ αργά. Γι' αυτό εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι έχουμε, είχαμε και το, το πρόβλημα των, της σκόνης, όμως ε, χρειαζόμαστε τις δομές αυτές ε, όσο να τον πιο γρήγορα. Ε, σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σας και να ξέρετε ότι θα έχετε την, όλη την υποστήριξη της Επιτροπής μας. Κύριος Κάνσεν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ και εγώ σας ευχαριστώ Υπουργέ και σας εύχομαι κάθε επιτυχία, ιδίως στην αρχή της Προεδρίας. Πιστεύω ότι θα πρέπει να πετύχετε σοβαρά αποτελέσματα. Μιλήσατε για την ολοκληρωμένη αλυσίδα υποστήριξης. Είμαι απόλυτα υποστη... Ε, ότι έχετε, το έχετε δίκιο. Όμως ε, υπάρχουν πολλά ντοσιέ τα οποία είναι αυτόνομα ε, για κάθε, και ανεξάρτητα και εξελίσσονται ανεξάρτητα για κάθε τρόπο μεταφοράς. Χρειαζόμαστε χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε τις μεταφορές ε, εναέριες, χερσαίες και θαλάσσιες σαν ένα ενιαίο σύστημα. Να έχουμε αυτό το όραμα μιας συνοπτικής ε, αντιμετώπισης. Τώρα, όσον αφορά τις, την, χρηματοδότηση, τα μέσα χρηματοδότησης, επιτρέψτε μου να επιμένω στο θέμα αυτό, στην εσωτερικοποίηση του κόστους, τα περιφερειακά ταμεία, τα άλλα κονδύλια του προϋπολογισμού, ο ορθολογισμός, η εκλογήκευση είναι ένα θέμα και σημαντικό. Αλλά όλοι λένε από τον παρόσο και κάτω ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί και ένα ειδικό ταμείο για τι τις για τα δίκτυα TEN, όχι μέσα στον κανονικό προϋπολογισμό, όπου θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε ε, χρηματοδότηση για κάθε ε, πρόγραμμα, για κάθε project. Αυτό είναι το θέμα στο οποίο πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας, ε, κύριε Πρόεδρε. Θα πρέπει να δούμε ότι ο χρόνος πιέζει και θα ήθελα να πω στον κύριο Κόζα ότι όλοι ε, οι επιβάτες, όλα τα δικαιώματα των επιβατών θα πρέπει να δυσοριστούν ανεξάρτητα από το μέσο ε, μεταφοράς. Έχει απόλυτο δίκαιο. Ο κύριος Λιμπεράτσικη για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα με ενδιαφέρον το πρόγραμμά σας, κύριε Υπουργέ. Πρέπει να σας πω ότι εξεπλάγιν ε, ήταν και πολύ ευχάριστη η έκπληξή μου γιατί θυμάμαι την παρουσίαση που έκανε ο Πρωθυπουργός στο Στρασβούργο. Από ό,τι κατάλαβα θα υπάρξει ένα καινούριο στοιχείο που αφορά τις, θαλάσσι, τις εσωτερικές ε, θαλάσσιες μεταφορές ε, και τον Δούναμι. Η πολιτική για το τι TNT και οι όμορες χώρες. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω την άποψή σα Θα υπάρξει κάποιο άνοιγμα προς την Ουκρανία ή στην Ρωσία, κάποια προσπάθεια έτσι ώστε να υπάρχει μια μεγαλύτερη συνοχή στις μεταφορές. Διότι είχαμε, μια, ε, είχαμε κάποιες εμπειρίες. Καταρχάς, ε, ε, είχαμε το ηφαίστειο που εξεράγει, τα αεροδρόμια που κλείσανε και δεν είχαμε καμία εναλλακτική λύση στην Ευρώπη. Τώρα το χειμώνα οι σιδηροδρομικές γραμμές κλείσανε στην Πολωνία, αλλά τα ίδια προβλήματα είχαμε και στην, στο Μένο Βασίλειο και σε άλλες χώρες. Επομένως, μήπως θα μπορούσαμε να σκεφτούμε νέα μοντέλα μεταφορών μετά την, την κρίση, μετά τα προβλήματα. Δηλαδή θα πρέπει να βρούμε και εναλλακτικού τρόπους. Ε, ε, αναφερθήκατε στην Ευρωβινιέτ και στο εξωτερικό κόστος και στον κανόνα ο χρήστης πληρώνει. Όμως, πόσα χρήματα μπορούν να πληρώνουν οι μεταφορικές εταιρείε έτσι ώστε να μην χρεοκοπήσουν από την άλλη, να μην χάσουν και την ανταγωνιστικότητά τους από την άλλη. Πιστεύω ότι φτάνουμε στα όρια. Και έχω την υποψία ότι τελικά δεν θα μπορέσουμε να αντέξουμε τον εξωτερικό ανταγωνισμό. Ευχαριστώ. Ja, vielen Dank, Herr Minister. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und ganz starke Nerven. In Ευχαριστώ, Υπουργέ. σα εύχομαι κάθε επιτυχία και ελπίζω να τα νεύρα σα να αντέχουν το επόμενο, να αντέξουν το επόμενο εξάμεινο. Είπατε, Υπουργέ, ότι οι περιβαλλοντικοί παράγοντε θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να ε, τις αγνοήσουμε, να τις παραμερίσουμε για οικονομικούς λόγους. Ολόκληρες περιοχές του Δούναβη κινδυνεύουν από να καταστραφούν λόγω των εγκαταστάσεων που δημιουργούνται εκεί. Γι' αυτό θα ήθελα, ε, Υπουργέ, προς Θεού, να μην υποκύψουμε στο κέρδος, στο άλογο κέρδος και στη χώρα μου, ο Δούναβης, ιδίω στην κάτω Βαβαρία, υπάρχουν, ε, δημιουργούνται Υπάρχουν πολλές ανησυχίες από τον τοπικό πληθυσμό λόγω των εγκαταστάσεων ε, στον Δούναβη που διευρύνονται. Λοιπόν, ε, μην αποφασίσουμε πράγματα χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας και τις ανησυχίες των του τοπικού πληθυσμού πρόεδρος. Έχω συμπεριλάβει και δύο άλλους ε, συναδέλφους γιατί ε, κάποιοι μίλησαν λιγότερο. Όμως ήθελα να πω ότι δεν μου αρέσει καθόλου το γεγονός ότι κάποιοι έρχονται στην αίθουσα αφού μιλήσει ο Υπουργό και μετά θέλουν να κάνουν και μια ερώτηση. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και προβλήματα, αλλά καλό θα είναι στο μέλλον, πριν ζητήσετε το λόγο, να έρθετε να ακούσετε τον Υπουργό κιόλα, κύριο κύριος Κράμερ. Σωστά, σωστά το είπατε κύριε Πρόεδρε. Λυπούμε. Συγγνώμη που έφτασα αργά, μου πρέπει να πάω και σε μια άλλη ε, συνεδρίαση και συζήτησα με την κυρία Λίχτεμπερκ που μου είπε ότι το θέμα που θα θίξω εγώ δεν έχει τεθεί ως, ερώτηση, ε, ερώτημα από άλλους συνεδρίους. Πιστεύετε κύριε Υπουργέ ότι μεταξύ των διαφόρων ειδών μεταφορών υπάρχει ε, σωστός ανταγωνισμό Δεδομένου ότι για τις οδικές ε, μεταφορές ε, δεν υποϊσχύουν παντού οι ίδιες ε, συνθήκες, για να αναφέρω ένα παράδειγμα τώρα, για το Δούναβι. Ο Δούναβης είναι ελκυστικός και για άλλους λόγους, όχι μόνο για την εσωτερική ναυσιπλοεία. Επίσης πρέπει να πω ότι υπάρχουν και πάρα πολύ ωραίε διαδρομές για να κάνει κανείς ποδήλατο. Θα πρέπει να προστατεύσουμε την ομορφιά της Σε Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ κυρία Υπουργέ. Σα δίνω 10 με 12 λεπτά για να απαντήσετε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πρώτη ερώτηση αφορούσε, αν δεν κάνω λάθος, τα δικαιώματα των επιβατών. Καλό θα ήταν να έχουμε ενιαίους αγώ... κανόνες για τα δικαιώματα των επιβατών σε όλη την Ευρώπη. Πρόσφατα συζητήσαμε τους κανόνες που πρέπει να ισχύουν τα δικαιώματα των επιβατών που ταξιδεύουν με λεωφορεία. Νομίζω ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να εναρμονίζουμε τους κανόνες. Δεν ξέρω. Όμως, τι πρέπει να γίνει με εναρμόνιση. Δεν ξέρω αν μπορούμε εδώ να έχουμε εναρμόνιση, αλλά ας έχουμε έστω μία περιορισμένη εμβέλεια συμφωνία, γιατί να έχουμε καθόλου συμφωνία. Αναφέρατε για τα λεωφορεία τα 250 χιλιόμετρα, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Ναι, θα έπρεπε οπωσδήποτε να γίνει λιγότερα. Εν πάση περιπτώσει. Δυστυχώς, οι δερμηνείς δεν ακούνε την κουβεντούλα που γίνεται στην αίθουσα. Εν πάση περιπτώσει, θα μεταφέρουμε το ερώτημά σας. Δεν ξέρω εάν αυτό είναι ένα θέμα που θα μπορέσει να συζητηθεί κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Για να απαντήσω στην κυρία Γκουρμάη. Το ερώτημα το οποίο αφορά τις ταχυδρομικές μεταφορές ε, θα το συζητήσει ο συνάδελφος ε, στην ε, Ήτρα, στην Επιτροπή Ήτρα αύριο. Η κρίση των αερομεταφορέων είναι ένα άλλο θέμα. Και εμείς έχουμε πρόβλημα. Και αν σας έλεγα θα το λύσουμε το πρόβλημα, θα μου λέγατε γιατί δεν ασχολείστε με το δικό σας αερομεταφορέα πρώτα παρά προσπαθείτε να λύσετε τα προβλήματα των αερομεταφορέων στην Ευρώπη πρώτα. Είναι πάρα πολύ, ε, πολλές οι πρωτοβουλίες και οι προτάσεις που έχει να παρουσιάσει για το θέμα αυτό η Επιτροπή και παρακολουθούμε ενδιαφέρον. Το Σίζαρ τώρα. Μπορώ να πω ότι πρόκειται για ένα θέμα πολύ σημαντικό για την ενιαία εσωτερική αγορά. Οι τιμές των εισιτηρίων, η στάχτη, είναι θέματα τα οποία θα συζητήσουμε στη διάσκεψη που θα λάβει χώρα το Μάρτιο και θα ακούσουμε και τις προτάσεις όλων των ενδιαφερομένων και εμπλεκομένων φορέων, των ενώσεων χριστών και θα τις λάβουμε υπόψη στις συζητήσεις. Τώρα, για την ε, σκόνη του ηφαιστείου, τι μπορούμε να κάνουμε. Βεβαίως, σε κάποιες χώρες της Ευρώπης με τα ταχεία τρένα, τα, ταχεία τρένα συγγνώμη, που έχετε κάτι μπορείτε να κάνετε, αλλά δεν είναι, συμβαίνει το ίδιο και με όλες τις χώρες της ε, κεντρικής και ανατολικής ε, Ευρώπης. Δεν είναι δυνατόν να αντικατασταθούν οι ενέργειες μεταφορές με σιδεροδρομικές, παρά το γεγονό ότι είναι ε, πιο φιλικές προς το περιβάλλον ίσως, αλλά δεν είναι πολλές φορές εξίσου φθηνές και γρήγορες. Ούτως ή άλλως τα ευρωπαϊκά συστήματα θα πρέπει να τα εναρμονίσουμε, αλλά να τα κάνουμε όσο πιο ανταγωνιστικά γίνεται. Όπως σας είπα, τα πάντα αλληλοεξαρτώνται στον τομέα των μεταφορών. Δεν μπορεί κανείς να προχωρήσει τον τομέα και να αφήσει κάποιον άλλο. Θα πρέπει σιγά σιγά σε όλους τους τομείς των μεταφορών να επιτυγχάνουμε πρόοδο. Και εμείς βασιζόμαστε στην πρόοδο που επέτυχε η Βελγική Προεδρία και ελπίζουμε ότι θα αφήσουμε και κάτι το θετικό για την επόμενη, την Πολωνική Προεδρία. Η Κομισιά και το Συμβούλιο συνεργάζονται. Κάθε Προεδρία βεβαίως μπορεί να εισαγάγει τις δικές προτεραιότητες, αλλά μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων της καθεμία Τώρα, η εσωτερική ναυσιπλοεία. Με τα TNTs βλέπουμε πώς μπορούμε να αναπτύξουμε διαφορούς διαδρόμους, διαφορά δίκτυα. Ε, μπορούμε να φτάσουμε μέχρι την ε, Μανία, την Ουκρανία. Θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε και ξέρουμε ότι πρέπει να είμαστε και στον τομέα των μεταφορών ανοιχτοί. Δεν μπορούμε να κάνουμε ένα οχυρό και για τις γραμμές εσωτερικής ναυσιπλοΐας στην Ευρώπη. Και θα πρέπει κάποιες συμφωνίες να τις επιτύχουμε και να τις διαπραγματευτούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και η Ουκρανία και η Μόσχα ξέρουν ότι πολλές φορές θα πρέπει να κάνουν συμφωνίες με όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα πρέπει να μιλάει με μία φωνή. Τώρα, η προστασία της περιοχής της Παραδουνάβιας και η προστασία του Δούναβη. Όταν μιλούμε για πράγματα, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, πάντα να προσπαθούμε να βρίσκουμε μία συμβαστική λύση. Η προστασία από πλημμύρες είναι εξίσου σημαντικό θέμα. Και θα πρέπει να προστατεύουμε τα συστήματα όλα στις ε, παραδουνάβιες περιοχές. Ξέρουμε ότι εξαιτία των κλιματικών αλλαγών έχουμε όλο και περισσότερες πλημμύρες και θα πρέπει να προσπαθούμε να προστατεύουμε τις περιοχές που θα μπορούσαν δυνητικά να υποφέρουν από αυτές τις πλημμύρες. Η κατάσταση στο είναι διαφορετική με την ε, εσωτερική ναυσιπλοεία από ότι το 70 ή το 80, κάποιες δεκαετίες πριν. Ακόμη και σε επίπεδο ε, κήτης του ποταμού θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν αλλαγές και θα πρέπει οι εμπειρογνώμονες σε θέματα περιβάλλοντος να μας συμβουλεύσουν και να μας πούνε τι είδους μέτρα θα πρέπει να λάβουμε χωρίς να καταστρέψουμε το Δούναβι και το φυσικό του περιβάλλον. Τώρα, μιλήσατε για το ΦΠΑ. Για τις, για τις αερομεταφορές, για ΦΠΑ στους αυτοκινητοδρόμους, δικές μεταφορές. υπάρχουν για τέτοιου είδους θέματα αντιφατικά και δύσκολα μεγάλες εντάσεις και διαφορές μεταξύ κρατών μελών. Και υπάρχουν θέματα τα οποία ποτέ κανείς δεν χειρίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο γιατί δημιουργούν πρόβλημα. Με την Ευρωβινιέτα πρέπει να πω ότι κάνουμε κάτι το πολύ καινοτόμο και καινούριο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα, Πόσο αυτό θα καταστήσει τον τομέα των μεταφορών πιο ανταγωνιστικό, πιστεύουμε ότι η Ευρώπη είναι μια ενιαία εσωτερική αγορά που πρέπει να έχει τους ίδιους ανταγωνιστικούς κανόνες για όρους. Πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί, αλλά να έχουμε τους ίδιους κανόνες και βεβαίω, όταν μιλούμε για λύση του προβλήματος δεν μιλάμε για λύση την οποία μπορούμε να επιφέρουμε σε έξι μήνες και να ζει για έξι μήνες. Αυτό που θα κάνουμε είναι κάτι το οποίο θα πρέπει μακροπρόθεσμα να αποτελέσει λύση. Έξι μήνες δεν είναι μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σκίσουμε με επιτυχία την Προεδρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ λέει ο πρόεδρος, ευχαριστούμε για την παρουσίαση που κάνατε και για τις απαντήσεις που δώσατε στις ερωτήσεις των μελών ε, της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ επίσης και τα μέλη της Επιτροπής για τις ερωτήσεις που έθεσαν ε, σαν Επιτροπή Μεταφορών και τουρισμού. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία το επόμενο εξάμεινο και περιμένουμε να σας ξαναδούμε τουλάχιστον προς το τέλος της Προεδρίας σας για να γίνει ένας απολογισμός του τι κάνατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας αφιερώσατε χρόνο και ήρθατε εδώ σήμερα. Okay, Συνάδελφοι, θα περιμένουμε λίγο. Πέντε ε, λεπτάκια, ούτω ώστε ο υπουργό και η αυλή του, επιτρέψτε μου να το πω, που συνήθω συνοδεύει του υπουργού, αποχωρήσουν από την αίθουσα.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 all the state secrets of Hungary there for us, yeah? <laughs> okay, colleagues, next item on the agenda. Συνάδελφοι, επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση της κυρίας Ερατσιάνη για τον ενιαίο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό χώρο. Δέμπορα, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως ξέρετε, μιλάμε εδώ για ένα θέμα για το οποίο ε, θα έχετε ε, σχετικά έγγραφα. Πρόκειται για την αναδιατύπωση τριών οδηγιών από το 2001 Θα ήθελα να σας πω ποια είναι τα κύρια στοιχεία της πρότασης που κάνει η Επιτροπή για την αναδιατύπωση. Να τα υποστηρίξω τα θέματα που πραγματεύει στην πρόταση της Επιτροπή και σας παρουσιάσω την έκθεσή μου. Στις προτάσεις Επιτροπής προβλέπεται αναδιατύπωση των τριών οδηγιών, κυρίως για την διασφάλιση της εποπτείας της αγοράς. Γι' αυτό προβλέπεται σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής κάποιος ανεξάρτητος διαχειριστής και άνοιγμα της αγοράς, πρόσβαση ε, στις διάφορες υπηρεσίες αδειοδότηση σιδεδρομικών επιχειρήσεων, ώστε γενικότερα να έχουμε άνοιγμα της αγοράς. Στην πρόταση Επιτροπής δεν αναφέρονται μόνο οι εθνικές αρχές διαχείρισης που πρέπει να είναι ανεξάρτητες, αλλά και διάφορα δίκτυα τα οποία θα μπορούσαν να χειριστούν θέματα ε, διασυνοριακά. Επίσης, προβλέπεται ένας ρυθμιστικός φορέας, μια ρυθμιστική ανεξάρτητη αρχή, Το δεύτερο θέμα αφορά την έλλειψη χρηματοδότησης που υπάρχει στον τομέα των σιδηροδρόμων, πράγμα το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το τόνισε πολλές φορές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, το λαμβάνει υπόψη και εμείς ε, προτείνουμε όπως η Επιτροπή να υπάρχουν νέες διατάξεις για να βελτιωθούν οι τα συστήματα χρηματοδότησης των σιδηροδρομικών ε, υποδομών. Και τα θέματα πρόσβασης σε διάφορες υπηρεσίες. Προβλέπονται λοιπόν διάφορα κίνητρα για την εγκατάσταση του εξοπλισμού ERTMS. Όλα αυτά τα θέματα επίσης αφορούν θέματα πρόσβασης σε διάφορες υπηρεσίες και εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης. Επίσης θα προβλέπεται διαχωρισμό διαχείριση υποδομής και λειτουργίας των μεταφορικών υπηρεσιών τα θέματα διαχείρισης της ε, υποδομής θα πρέπει να παραμείνουν θέματα αρμοδιότητας των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολλές φορές είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει πραγματική ανεξαρτησία μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών. Και εγώ είμαι υπέρ αυτού του διαχωρισμού. Και το αναφέραμε και στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου τον Ιούνιο του 2010. Το προσφέρω βέβαια προς συζήτηση το θέμα αυτό, γιατί πιστεύω ότι θα πρέπει να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειε και να βρούμε ποια είναι η καλύτερη δυνατή λύση. Ένα τελευταίο θέμα, το οποίο θα ήθελα να υπογραμμίσω, συνδέεται με ένα θέμα το οποίο είναι πιο διοικητικό και τεχνικό, θα έλεγα. Σχετίζονται με τα παραρτήματα τα οποία έχουν επισυνεχθεί στην πρόταση της Κομισιόν. Ξέρετε ότι η Κομισιόν για λόγους ευελιξίας και ε, προσαρμογής των προβλέψεων ε, στις ε, διάφορες πολιτικές και νομικές εξελίξεις μπορεί να τροποποιήσει τα παραρτήματα αυτά. Όμως πρόκειται για πάρα πολύ σημαντικά παραρτήματα τα οποία συνδέονται με την πρόταση οδηγίας. Επομένως, εάν τροποποιηθούν τα παραρτήματα θα θυγούν σημαντικές, σημαντικά στοιχεία της οδηγίας. Γι' αυτό θα πρέπει να αξιολογήσουμε την σημασία κάθε επιμέρους παραρτήματος για να δούμε κατά πόσον το περιεχόμενο του παραρτήματος αυτό, αυτού μας, ε, ε, μας αναγκάζει να ε, χρησιμοποιήσουμε μάλλον για να δούμε ποιο τρόπο αλλαγή θα χρησιμοποιήσουμε, θα υιοθετήσουμε. Βέβαια καταλαβαίνω ότι χρειάζεται να γίνει μια συζήτηση ε, και είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Σερακιάνη. Πριν ε, προχωρήσουμε να πω ότι έχουμε ε, μεγάλο κατάλογο ομιλητών. Μιλάμε για ένα αρχικό κείμενο, έτσι, να το επενθυμίσω αυτό, δεν είναι το σχέδιο, οδηγίες, ε, το σχέδιο έκθεσης. Επομένως, έχουμε 45 λεπτά στη διάθεσή μας για να το, να το ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό. Έχω πολλούς ομιλητές. Θα ξεκινήσω με τους σκιώδεις. Οι σκιώδεις ε, τρία λεπτά και οι υπόλοιποι δύο. Ο κύριος Κούνα από το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κυρία Σερακιάνη, για το έγγραφο αυτό. Ευχαριστώ την Κομισιό που κάνει, έκανε αυτή την πρόταση για την ε, οδηγία που αλλάζει, αν θέλετε, που τροποποιεί το, που αναδιατυπώνει ε, συγγνώμη, όλο το πακέτο του ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου Έχουμε συζητήσει τα άλλα θέματα για, τους, ε, για, τον, ε, για τις ενέργειες και τις χερσαίες μεταφορές. Εδώ στο σιδηρόδρομο ε, αντιμετωπίζουμε μεγάλα προβλήματα. Και γι' αυτό νομίζω ότι εδώ πρέπει να θέσουμε πάρα πολύ συγκεκριμένου όρους για το πώς θα πρέπει να λειτουργεί το management, η διαχείριση κτλ. Αν θα υπάρχει εποπτικό συμβούλιο ή συγκεκριμένη εποπτική αρχή κτλ. Και θα πρέπει να υπάρχει σαφήνεια, ακρίβεια και διαφάνεια και όσον αφορά τις, ε, των λογιστικών βιβλίων αν θέλετε στο συνδρομό και επίσης αυτό επηρεάζει και τις τιμές και κυρία Σερατσάνη μιλήστε για την ε, ε για την αριθμιστική κανονιστική αρχή Πρε, όντως πρέπει να υπάρχει ε, μια τέτοια κανονιστική ρυθμιστική αρχή αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να υπάρχει και ένας επόπτης, μια εποπτική αρχή και μια συντονιστική αρχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο διαφορετικά δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα πράγματα Κάποιος πρέπει να κάνει το συντονισμό, κάποιος πρέπει να επιβλέπει τα πράγματα αυτά διαφορετικά. Δεν υπάρχουν, ε, δεν θα κάνουμε τίποτα. Επί, κατά τα άλλα, συμφωνούμε ότι και ότι στο επίπεδο της ασφάλειας ε, πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες θα πρέπει επίσης να καθίσουμε να συζητήσουμε ε, ποιες είναι οι περιπτώσεις κατά τις οποίες α, ε, κατά τις επειδή η υποδομή δεν το επιτρέπει μπορούμε να προσθέσουμε αν θέλετε χωρητικότητες δυναμικό ε, και μία τέτοια περίπτωση είναι το στερικό το κέντρο των μεγάλων πόλων είτε είναι το Παρίσι είτε είναι το Βερολίνο ας πούμε εδώ υπάρχουν προβλήματα που πρέπει να μελετηθούν σε βάθος από εκεί και πέρα βέβαια η Κομισιόν Κομισιόν ε, ξεκίνησε μία ε, διαδικασία, έδωσε κάποιες εξουσίες αν θέλετε ε, Τώρα το θέμα είναι πώς θα εφαρμόσουμε εμείς αυτά που λέει η Κομισιόν, αλλά έχουμε από πού να ξεκινήσουμε. Από εκεί και πέρα βεβαίως πρέπει να δούμε και τα, την διαλειτουργικότητα και τις διασυνοριακές ε, Παραβάσει και καταγγελίες συμβάσεων. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς που δίνετε το λόγο, αλλά και την εισηγήτρια για τη δουλειά που έκανε είναι πράγματι σημαντικό να προσθέσουμε πολλά πράγματα ε, για να προ, αν θέλουμε να προωθήσουμε το σιδηροδρομικό ο, τις σιδηροδρομικές μεταφορές πρώτα πρώτα σε πολλές χώρες δεν υπάρχει πραγματική ρυθμιστική αρχή και εποπτική αρχή και τα λοιπά δεύτερο κυρίες και κύριοι, δεν έχει ανοίξει αγορά τελικά στην Ευρώπη. Σε κάποια κράτη-μέλη η κατάσταση είναι χειρό, χειρότερη από άλλες χώρες. Παράδειγμα, η Ισπανία. Μόνο 4% των συνολικών μεταφορών γίνονται με το σιδηρόδρομο βλέπουμε να ακολουθείτε και να υπάρχουν τάσεις τελείως αντίθετες από αυτές που θα έπρεπε να υπάρχουν. Εκ μέρους της πολιτικής μου ομάδας ε, θα ήθελα να πω ότι ε, ε, χαιρετίζουμε μερικά πράγματα που λέγονται στην έκθεση κυρία Σερατζάνη, απ' την άλλη με, επιμένουμε όμως σε μια ισχυρή ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή που θα εξασφαλίζει και ε, δίκαιο ανταγωνισμό και καλό συντονισμό και καλή, καλό άνοιγμα της αγοράς. Και εδώ είναι δύσκολο να προχωρήσουμε. Πρέπει να άρουμε όλα τα πιθανά φράγματα που υπάρχουν και θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε <coughs> να ε, εξασφαλίσουμε ότι τα κράτη-μέλη ε, θεσπίζουν και αυτά ε, ρυθμιστικές κανονιστικές αρχές στο εσωτερικό τους με ικανή χρηματοδότηση και ικανές αρμοδιότητες. Αυτές οι ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές θα έπρεπε ήδη να υπάρχουν τώρα στα κράτη-μέλη αλλά περμέναμε 10 χρόνια και αυτό δεν έχει ακόμη γίνει. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει κάτι να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να υπάρχει και εποπτεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο να η εποπτεία των, ε, αυτών των αρχών για να μπορέσουν τα πράγματα να προχωρήσουν. να δημιουργήσουμε, ίσως θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε και μια ειδική, ένα ειδικό τμήμα στην ε, ε, γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού ή ένα, μια ειδική αρχή, δεν ξέρω, σε ευρωπαϊκό επίπεδο που να αναλάβει όλη αυτή τη δουλειά που πρέπει που είναι απαραίτητο να γίνει. Θα μπορούσαμε να κάνουμε και μια μελέτη για το unbundling, που όπου θα περιγράφεται η κατάσταση σε όλα τα κράτη-μέλη και θα, προτείνουν, θα γίνονται και προτάσεις. Τα Η μελέτη αυτή θα πρέπει να αναφέρεται λοιπόν σε όλες τις επιμέρους ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών να μας λέει πώς είναι οργανωμένες, τι, τι κάνουν και Βεβαίω είναι πολύ σημαντικό να μελετηθεί και το θέμα του unbundling, αλλά ε, η μελέτη του unbundling δεν θα πρέπει να μας ε, από προσανατολίση από την προσπάθεια αναδιατύπωση, από την αναδιατύπωση που προτείνει εδώ τώρα η Κομισιόν. Με αυτό συμφωνούμε. Απλώς θέλουμε να πιέσουμε για να πάμε πιο πέρα από αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι, αν ακολουθήσετε όλο αυτό το παράδειγμα δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Ο κύριος Κράμερ όταν μεταρρυθμίζαμε τα του σιδηροδρόμου πριν από 15 χρόνια στη Γερμανία πιστεύαμε ότι θα πρέπει θα πρέπει να α, γίνει διάκριση και διαχωρισμός μεταξύ του δικτύου και των τη επιχείρηση, αν θέλετε σιδηρόδρομο. Εγώ συνεχίζω να την πιστεύω. Α, αυτή... Ε, Ε, εγώ συνεχίζω να πιστεύω ότι πρέπει να είναι κριτήριο αυτό ο διαχωρισμός δικτύου και επιχείρησης παρόλο που δεν είναι το μόνο αλλά τέλος πάντων βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη που αυτό το διαχωρισμό τον, ε, διαχωρισμό τον έχουν κάνει θρησκεία είναι οι τελευταίοι αυστηροί εθνικιστές αν μπορώ να το πω έτσι. Εν πάση περιπτώσει, εδώ και πολύ καιρό γίνεται προσπάθεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να ε, οργανωθούν να συντονιστούν ορισμένα πράγματα. Υπάρχουν τα, αλλά δεν βλέπουμε να γίνεται μεγάλη πρόοδος. Και αν δούμε στις διάφορες χώρες τι γίνεται με τις ρυθμιστικές αρχές, βλέπουμε ότι υπάρχουν ρυθμιστικές αρχές που παίρνουν αποφάσεις πραγματικές μέσα σε 14, σε ένα 15 θήμερο και άλλες οι οποίες περιμένουν χρόνια. Είναι πάρα πολύ διαφορετικά τα πράγματα στις διάφορες χώρες και η κατανομή των σλότς, η πρόσβαση στα διάφορα σλότς είναι μεγάλη υπόθεση αυτό και υπάρχουν και τρίκ και κόλπα που βλέπουμε στα διάφορα κράτη-μέλη και άμα ε, έχουμε μια χώρα που από 400 σλότς πέφτει στα 70 και ε, λέει μετά αν δεν έχουμε χώρο, τέρμα, δεν γίνεται, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα». Με κοροϊδεύει τον κόσμο. Αν θέλουμε να προχωρήσουμε το σιδηρόδρομο σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να κάνουμε κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε και αυτά που περιγράφονται εδώ αλλά θα πρέπει να γίνουν και πολλά πράγματα σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να γίνουν, υπάρχουν πραγματικές ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές, να, ε, ε, να υπάρχει ανεξαρτησία, να υπάρχει αποτελεσματικότητα και βεβαίως δεν λέω να υπάρχει και η εποπτεία και ο συντονισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά αν δεν κάνουν οι χώρες κάτι, τι, αν δεν νοικοκυρευτούν τα πράγματα σε όλες τις χώρες μέλη, δεν νομίζω ότι κάνουμε τίποτα. Το κριτήριο του διαχωρισμού δικτύου και επιχείρηση που λέγαμε στην αρχή ε, είναι κριτήριο βεβαίως αλλά υπάρχουν χώρες όπου ο διαχωρισμός αυτός είναι πλήρης αλλά δεν προχωράει τίποτα. Εδώ παίζουν άλλα πράγματα ρόλο. Η διαφάνεια παραδείγματος χάρη. Ευχαριστώ πολύ, πολύ Ζέλερ τρία λεπτά. Λοιπόν, θα ήθελα να σχολιάσω αυτά που ελέγχθησαν. Ο ένα η μία και μόνη ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή που αναφέρθηκε και από άλλους. Είναι απαραίτητη ε, η Rail Agency που υπάρχει αυτή τη στιγμή δεν έχει τις απαραίτητες αρμοδιότητες και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ίσως πρέπει να, ε, όπως και στις τηλεπικοινωνίες, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές να αυτονομηθούν και να γίνουν διαφανέστερες αλλά από εκεί και πέρα ίσως θα πρέπει να υποπτεύονται από κάποια ευρωπαϊκή αρχή τώρα για το unbundling Αυτό όμως, αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο όμως σχετίζεται και με το άνοιγμα των αγορών. Ε, αν τελικά καταλήξουμε σε μία μονομαχία μεταξύ δύο μεγάλων ε, επιχειρήσεων στην Ευρώπη για το ποιο θα έχει το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς τα πράγματα για μένα θα είναι τραγικά ε, δεν πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο εμείς θέλουμε πραγματικά ανοιχτή αγορά ελεύθερη αγορά στις χώρες της Βαλτικής έχουμε ένα είδος ειδική τροχιάς. Έχουμε συζητήσει με ε, τους αρμόδιους και έχουμε καταφέρει και Ξέρουμε ότι οι τροχές ε, στην Ευρώπη είναι διαφορετικές από ό,τι εμάς. Σε εμά λοιπόν υπάρχει διαλειτουργικότητα με τη Ρωσία, αλλά όχι με την υπόλοιπη Ευρώπη. Προσκαλούμε τους Ευρωπαίους να έρθουν στη χώρα μας. είναι σημαντικά και τέτοιου είδους τεχνικά προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ. οι σιδηρόδρομοι έχουν και μια κοινοφελή πτυχή. Δεν ε, μεταφέρουν μονάχα εμπορεύματα, μεταφέρουν και ανθρώπους που πάνε στη δουλειά τους. Και με αυτή την έννοια ο εθνικός χαρακτήρας των σιδηροδρόμων είναι δεδομένος. Υπάρχουν δικαιώματα των επιβατών που πρέπει να προστατεύσει το κράτος μέλος. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις μεταφορές με την έννοια των εμπορευματικών μεταφορών, θα... εκεί ε, δίνονται άδειες, εκεί ε, δίνονται άδειε και σε επιχειρήσεις που δεν προέρχονται καν από τον σιδηροδρομικό χώρο και άρα δεν έχουν μεγάλη πήρα που δεν ήταν πάντα κρατικές ε, ή δεν είναι κρατικές και εδώ δημιουργούνται προβλήματα όσον αφορά τις θέσεις απασχόλησης. Άνοιγμα των αγορών ζητιέται, ωραία, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να, υπάρχουν και έντονοι και αυστηροί κανόνες που να τηρούνται. Αυτά, αυτό, αυτά όμως όλα είναι θέμα των κοινοβουλίων. Ε, τα κοινοβούλια θα πρέπει να αποφασίσουν τι θα γίνει και θα πρέπει να δουν βεβαίως ε, είναι δική τους δουλειά να ε, δουν τι γίνεται με τις ρυθμιστικές και κανονιστικές αρχές και είναι δική τους δουλειά να δουν και τι γίνεται με τις υποδομές. Στο παράρτημα 8, στο σημείο 9, αυτό που αναφέρεται για μένα είναι κακό για τις ελάχιστες υπηρεσίες, για τα ελάχιστα προότυπα κτλ. Είναι λάθος. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι θέμα της Ευρώπης να καταπολεμά τις απεργίες ή να αγωνίζεται κατά των απεργών από εκεί και πέρα και για τις αμοιβέ. Ε, ε, αυτά που αναφέρονται εδώ είναι λάθος. Συνάδελφοι, έχουμε ένα κατάλογο 14 ομιλητών. Είχαμε 15, αλλά η κυρία Ντουράν πάρα πολύ ευγενικά αποσύρθηκε. Λοιπόν, 14, 14 ομιλητέ. Κομισιόν και κυρία Σερακιάνη στο τέλος. Επομένω, σεβαστείτε τα δύο λεπτά. Συμφωνώ ότι είναι πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον το θέμα. Όμω, πρόκειται για ένα προκατακτικό έγγραφο. Δεν είναι το σχέδιο έκθεση. Λοιπόν, Όλα πρέπει να λεχθούν, αλλά δεν πρέπει να τα πούνε όλοι όλα. Επομένως, ξέρω ότι θα ακούσουμε πολλές επαναλήψεις, αλλά τι να κάνουμε, ο άνθρωπος πάντα λυπίζει. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και την εισηγήτρια, ευχαριστούμε και την Κομισιόν για τις προτάσεις. Θα θέλαμε να προσεγγίσουμε το θέμα όχι με δογματικό τρόπο θα, νομίζω ότι θα πρέπει πρώτα πρώτα να, δω, να αναρωτηθούμε τι, ποιοι είναι οι στόχοι μας και αν μπορούν να επιτευχθούν. Άνοιγμα της αγοράς δεν είναι αυτός σκοπός αυτό. Ε, το άνοιγμα της αγοράς είναι καλό άμα βελτιώνεται μα με το άνοιγμα η υπηρεσία που παρέχεται. Και αν δούμε τώρα την κατάσταση έτσι όπως είναι εδώ θα πρέπει να έχουμε αμφιβολίες. Δεύτερον, τα, ποια είναι τα μέσα που ε, ε, είχαμε κατά νου. Ε, είπαμε ε, ρυθμιστική αρχή Είχαμε πει τότε ρυθμιστική αρχή που επιβάλλει ορισμένου κανόνε κτλ. Είχαμε τρει στόχου σχετικά με αυτό. Κανένα δεν επετεύθη. Αποτύχαμε. Τώρα λοιπόν εδώ τι προσπαθούμε να κάνουμε θέλουμε να βελτιώσουμε τα πράγματα όχι πρώτα σε εθνικό επίπεδο και μετά σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά κατευθείαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν ξέρω αν μπορούμε να το κάνουμε επίσης αν ε, προσπαθήσουμε να ρυθμίσουμε τα πράγματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο τι θα γίνει με τη χρηματοδότηση τι τέλη θα υπάρχουν τι θα γίνει με την υποδομή και δυστυχώς ο έλεγχος, ο οποίος είναι το α και το ω. Αγαπητοί, αν αύριο θέλουμε μια ανοιχτή αγορά με υγιείς κανόνες ανταγωνισμού, είναι απαραίτητο να έχουμε και έναν αυστηρό κριτή, ε, αυστηρό έλεγχο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και εδώ Πραγματικά θα πρέπει να κάνουμε διάκριση μεταξύ του, οργανισμού της Rail Agency και της ρυθμιστικής αρχής του Regulator που είναι τελείως άλλο πράγμα. είμαστε θετικοί για την προώθηση των σιδηροδρόμων. Από την άλλη μεριά θέλουμε να είμαστε και ρεαλιστές και δεν βλέπουμε ε, να γίνονται πολλά πράγματα εύκολα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το έγγραφο αυτό. Μου φαίνεται ότι το μέλλον της αγοράς των σιδηροδρόμων δεν θα πρέπει να υπακούει μόνο στους αγ κανόνες της αγοράς. Είναι σημαντικό το θέμα και των υποδομών και της διαλειτουργικότητας. Αυτά τα τρία στοιχεία θα πρέπει να τα λάβουμε σοβαρά υπόψη. Όσον αφορά τη λειτουργία της αγοράς, πιστεύω ότι όλοι είμαστε υπέρ του ανοίγματο που πρέπει να γίνει με επιτυχία. Και σοβαρά, ένα από τα βασικά στοιχεία είναι το θέμα της ε, ρυθμιστικής αρχής που θέλει να ενισχύσει την εκθεσή της η συγγεντρία. Μιλά ακόμη και για ένα δίκτυο ρυθμιστικών αρχών. Θα πρέπει να είμαστε ακόμη πιο φιλόδοξοι, να κάνουμε κάτι το οποίο να είναι πραγματικά ως φορέας, ως αρχή ευρωπαϊκό και να λειτουργεί σωστά. Στο θέμα του διαχωρισμού τώρα, θα πρέπει να δούμε τελικά τι θέλουμε να επιτύχουμε. Θέλουμε να έχουμε ίσους όρους, να μην έχουμε διακρίσεις, να έχουμε διαφάνεια, να έχουμε την ίδια ε, τιμή, αν θέλετε, για όλους. Θα θέλαμε να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα αυτό. Η συγγήτρια πρέπει να πάρουμε τελική μας απόφαση. Επίσης, θα θέλαμε να ξέρουμε για τα θέματα αδειοδότησης περισσότερα πράγματα. Επίσης υπάρχουν διαφορές μεταξύ των διαφορών των μελών, διότι δεν υπάρχει τίποτε το ενιαίο, το ευρωπαϊκό, αν θέλετε. Κάτι άλλο που θέλω να προσθέσω είναι το θέμα του κόστους των έργων υποδομής. Οι κανόνες που ισχύουν και τα πρότυπα είναι τόσο διαφορετικά από τη μία χώρα στην άλλη που για να κάνουμε ενοποίηση θα πρέπει να μελετήσουμε πολύ ακόμη το θέμα. Κυρία Μάιστερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλουμε πράγματι με έναν ε, ενιαίο σιδηροδρομικό χώρο στην Ευρώπη. Δεν τα προσπαθούμε εδώ και χρόνια, δεν τα καταφέραμε. Ε, είναι σημαντικό είναι παράξενο βέβαια γιατί συμφωνώ και πάλι με τον Μιχάλ εδώ θα μπορούσα και να κάνω πολλά πράγματα εάν ε, ήμουνα σίγουρη για κάποια αποτελέσματα αλλά δεν μπορώ, μπορώ να είμαι σίγουρη για τα αποτελέσματα διότι οι προσπάθειες που έγιναν μέχρι τώρα δεν απέδωσαν καρπούς λυπάμαι Ο κύριος Ρίκη Εν συντομία κύριε Πρόεδρε ευχαριστώ καταρχάς να συγχαρώ την κυρία Σερακιάνη για την δουλειά της για τη θέση της ε, που θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Όλοι είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, δεν πρόκειται να κάνω έναν κατάλογο όλων των θεμάτων, αλλά να πω ότι όλοι λένε ότι θα πρέπει να ανοίξουμε με έναν ε, ισορροπημένο, συνδεδεμένο, αποτελεσματικό τρόπο το σιδηροδρομικό δίκτυο, αλλά το προηγούμενο κείμενο οδήγησε 13 χώρες ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Προβληματικό αυτό. Δεύτερο, ε, το επίπεδο των επενδύσεων συνδέεται με τη λειτουργικότητα του δικτύου. Εάν ε, έπρεπε ε, με τη μεταφορά, όταν γίνεται μια μεταφορά με φορτηγά ε, σε κάθε, σε κάθε διάβαση των συνόρων να πρέπει να αλλάζω κινητήρα, να αλλάζω φορτηγό, να αλλάζω οδηγό, το πράγμα δεν λειτουργεί. Επομένως, θα συμφωνώ με τη θέση της συγγήτριας εδώ. Επίσης να πούμε ότι συμφωνούμε με το, σκοπό, με το στόχο, αλλά ο καθένας έχει τις δικές του απόψεις, το πράγμα τα επίσης δεν θα προχωρήσουμε. Εάν θέλουμε να έχουμε ένα ανοιχτό, διάφανο και ανταγωνιστικό ε, σύστημα και αγορά, θα πρέπει τα πάντα να γίνουν ταυτόχρονα. Δεν πρέπει να γίνεται πότε το ένα, πότε το άλλο κτλ. Δεν πρέπει να προχωρήσουμε έτσι. Όλα τα μέτρα θα πρέπει να τα ε, λάβουμε ταυτόχρονα και όλοι θέλουν να υπάρχει ένας Ευρωπαίος ρυθμιστής με αρμοδιότητες, με εξουσίες. Ε, θέλουμε να υπάρχουν αν θα πρέπει να ανοίξουμε τι αγορέ, προφανώ πρέπει να ανοίξουμε τις αγορές. Πρέπει να ανοίξουμε τις αγορέ σε περιφερειακό πεδίο, Προφανώ. Δεν καταλαβαίνω την θέση που λέει, συμφωνούμε όλοι όσον αφορά το στόχο, αλλά από εκεί και πέρα ε, ο καθένας επιλέγει κάποια μέτρα που τον βολεύουν. Όχι, θα πρέπει όλα να ιδρυθούν ταυτόχρονα και θα πρέπει να υπάρχει συνεχής έλεγχος. Και επίση θα πρέπει να ξεκινήσει και αυτό το τρένο πλέον των ε, ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων. Ε, θα πρέπει τα πάντα να τεθούν επιτάπητος, να τα διαλύσουμε και να τα ξαναφτιάξουμε όλα μαζί. Γιατί αν δεν το κάνει το κοινοβούλιο, δεν το κάνει κανείς, ούτε καν η Κομισιό, η οποία ε, μας υπέβαλε ένα, ένα έργο το οποίο δεν είναι και ιδιαίτερα ε, αποτελεσματικό. Κύριο Κόλτσεκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή των συναδέλφων σε κάποια θέματα. Το συνδρομικό πακέτο δεν, δεν έχει εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη-μέλη. Μπορούμε να λέμε συνέχεια για το άνοιγμα της αγοράς κτλ. Αλλά γιατί από τα, 20, 25 κράτη-μέλη τα οποία έχουν σιδηροδρόμους δεν ε, υπήρξαν ε, αποτελεσματικά βήματα για την υλοποίηση ε, του συνδρομικού πακέτου. Θα ήθελα μία εξήγηση. Επίσης, πιο αποτελεσματικό είναι τα, το σύστημα RTMS, τεχνικής συμβατότητας Έχουμε διάφορα, διάφορες, διάφορους κινητήρες, ε, διάφορες μηχανές υδροδρομικές ε, που είναι συμβατές μεταξύ τους, όμως δεν έχουμε συμβατούς κανονισμούς ασφάλειας. Μπορούμε να έχουμε ένα πολύ καλό ρυθμιστή, αλλά εάν δεν θέλουν να συμμορφωθούν τα κράτη-μέλη, δεν θα πετύχουμε. Επίσης πρέπει να σας πω ότι στο παρελθόν μπορούσαμε να ταξιδέψουμε στην Ευρώπη σιδηροδρομικά χωρίς μεγάλη γραφειοκρατία, πολύ λιγότερη από ό,τι τώρα. Επομένως, πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους σιδηροδρόμους. Η αναδιατύπωση του πρώτου σιδηροδρομικού πακέτου δεν θα βοηθήσει, ανεξάρτητα αν υπάρχει καλή θέληση ή όχι. Äh, äh, και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω συνάδελφο Σερακιάνη για το έγγραφό της και νομίζω ότι κατέστη πλέον σαφές αγαπητοί συνάδελφοι για ε, σε όλους ότι εκείνο που θέλουμε να κάνουμε είναι να προχωρήσουμε σε ένα ενιαίο χώρο δίχως διακρίσεις. Βεβαίω το το unbundling, οι ρυθμιστικές αρχές, η ανάγκη επιβολής κανόνων και ρυθμίσεων είναι τα κύρια θέματα τα οποία ε, συζητούνται. Ήδη όμως υπάρχουν κάποια ε, πράγματα που εφαρμόζονται. Υπάρχει μια δομή holding η οποία α, δεν είναι κακή. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Και θα ήθελα να προτείνω μια συμβιβαστική λύση. Να ε, εστιάσουμε πρώτα-πρώτα την προσοχή μας στους ε, αυτούς που διαχειρίζονται την υποδομή και αν και εφόσον καταλήξουμε σε ένα πλουραλιστικό σύστημα εκεί για την υποδομή τότε πραγματικά όλα τα άλλα θα βρουν τη θέση τους και θα υπάρχει σωστό ε, ανταγωνισμός και θα υπάρχει και διαφάνεια και από εκεί και πέρα θα <coughs> ήθελα να προτείνω να ενισχύσουμε και τις ε, εθνικές ρυθμιστικές αρχές οι οποίες έχουν να λύσουν, θα πρέπει να λύνουν τα εσωτερικά προβλήματα αλλά και ε, σε συνεργασία ε, και προβλήματα ε, διασυνοριακά κτλ. Αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε μια Ευρωπαϊκή Αρχή, αλλά θα πρέπει να ισχύσει εδώ η αρχή της επικουρικότητας. Ε, ε, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Ένα σημείο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να έχουμε μία δήλωση, μία διευκρίνηση από τις ε, κανονιστικές αρχές Επομένως όλοι όσοι εργάζονται στο σιδηρόδρομο να ξέρουν τι ακριβώς ισχύει. Μία ερώτηση προς την Επιτροπή. Ένα από τα θέματα είναι η αποδέσμευση, το unbundling. Η Κομισιό έχει υποβάλει διάφορα έχει ξεκινήσει μάλλον κάποιες ε, διαδικασίες εναντίον των κρατών μελών. Εδώ στην επαναδιατύπωση της οδηγίας του πακέτου θα ε, ρυθμίσουμε τα θέματα της αποδέσμευσης ή όχι. Η θα πρέπει να, να δούμε τι, τι ακριβώς ε, μέλη γενέστε, διότι σε κάποια στιγμή θα πρέπει να προχωρήσουμε σε αναδιατύπωση αναδιατύπωσης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια που με σπέβαλε το κείμενο αυτό είναι πολύ καλό που γίνεται η συζήτηση αυτή και ήδη συμφωνώ με πολλά από αυτά που ελέγχθησαν ιδιαίτερα για τις ρυθμιστικές αρχές ενίσχυση των εθνικών αρχών και ύπαρξη μιας Ευρωπαϊκής Επιτροπή ε, Εποπτικής Αρχής ε, Τρόπων την Συντονιστικής ε, άρθρο 55 κτλ δεν ε, Έχω τώρα για, την, για τις υποδομές που αναφέρονται και την, το άνοιγμα της το, το ότι δεν μπόρεσαν να ανοίξουν οι αγορές είναι, οφείλεται κατά την άποψή μου στη, σε τεχνικά προβλήματα και έλλειψη διολειτουργικότητας ε, δεν νομίζω ότι ο ότι δεν μπορούμε πάντως να κάνουμε κάποια πράγματα εδώ. Συμφωνώ με πολλούς που μίλησαν για το θέμα αυτό. Ενίσχυση διαλειτουργικότητας και τη εξασφάλιση τεχνικής διαλειτουργικότητας. Εκείνο το οποίο δεν αναφέρεται εδώ καθόλου είναι τελικά το προσωπικό. Είναι οι εργαζόμενοι και νομίζω ότι δεν είναι σωστό αυτό. Δεν νομίζω ότι πιστεύει κανείς ότι δεν χρειάζεται το προσωπικό για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις μετατροπές αυτές τις οποίες θέλουμε να κάνουμε. Άρα θα πρέπει να προσέξουμε περισσότερο το προσωπικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ και την Τέμπορα για τη δουλειά που έκανε. Πιστεύω ότι το έγγραφο αυτό εργασία είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό είναι ένα φάκελο, ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να τον ε, προσέξουμε έτσι ώστε να μην χρειαστεί να κάνουμε μια επαναδιατύπωση στο μέλλον τη επαναδιατύπωση. Είπαμε ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο ανταγωνιστικό και στο κράτο και ανάμεσα στα κράτη. Ε, ούτως ή άλλως ε, μιλάμε ε, για ανταγωνιστική, αντιγωνιστικές αεροδρομικές μεταφορές για, μόνο για τους επιβάτες. Εδώ μιλάμε για ανταγωνιστικότητα, σήμερα μιλάμε για ελεύθερη αγορά κτλ. Γι' αυτό θα πρέπει να ανοίξουμε ε, Του σιδηροδρόμου, τουλάχιστον στι εθνικέ μεταφορέ και σε περιφερειακό επίπεδο βέβαια, που θεωρώ ότι είναι απαραίτητο, αλλά ε, και πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνουν βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Για να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζεται ο Ευρωπαίος ρυθμιστής, διότι η κατάσταση αντιμετωπίζεται από μία πηγή μόνο, από μία οπτική γωνία από την Ευρώπη. Επίσης θα πρέπει να διευρύνουμε τα θέματα... Ε, ασφάλειας αλλά και τυποποίηση ε, και έγκρισης ε, από πλευράς ε, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας. Τώρα όσον αφορά το unbundling αφορά, πρέπει να αφορά, αναφορά τις δραστηριότητες, όχι την ιδιοκτησία αν θέλετε, όχι το, τα υλικά. Υπάρχει, έγινε μια μελέτη νομίζω και θα πρέπει να, να δούμε τη μελέτη αυτή, γιατί θα πρέπει να κατανοήσουμε πώς οργανώνεται αυτή η πρωτοβουλία. Για μένα αυτό που μου είναι ενδιαφέρον είναι η... Θα πρέπει να ε, τα προϊόντα να λειτουργούν και να κυκλοφορούν ελεύθερα στην αγορά. Για μένα αυτό έχει σημασία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για, αυτή την, ε, για αυτό το τόσο ενδιαφέρον έγγραφο εργασία. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει αυτό το πακέτο το σιδηροδρομικό, ο τομέας ε, είναι κατακερματισμένος και μη ανταγωνιστικό. Οι επιβάτες, ε, οι υπεπολίτε δεν μπορούν να υποφεληθούν από τον κοινό σιδηροδρομικό χώρο. Η ίδια κατάσταση επικρατεί και στη μεταφορά των ε, εμπορευμάτων. Σε πολλές περιπτώσεις το θέμα της χρηματοδότησης δεν ήταν το μοναδικό πρόβλημα. Η έλλειψη πολιτικής ε, θέλησης στην εκπόνηση ε, υπερεθνικών προγραμμάτων είναι επίσης ένα σημαντικός παράγοντας. Πρέπει να εξασφαλίσουμε μια σωστή χρηματοδότηση για τις νομικές υποδομές. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να έχουν ε, τις, ε, τη χρηματοδότηση για την υλοποίηση των ε, project, διαφορών project εγκαίρως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η Κομισιόν να παίξει έναν ενεργό ρόλο στον έλεγχο και στην εφαρμογή των project που προβλέπονται σε εθνικό επίπεδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Φιντάνσα. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Σερακιάνη για αυτή την πρώτη παρουσίαση και στο κείμενο της Κομισιόν μπορούμε να εντοπίσουμε κάποια στοιχεία τα οποία μπορούμε να πλουστεύσουμε αλλά χρειάζεται κουράγιο κυρίως αναφορά αφορά το άνοιγμα της αγοράς και της ε, φιλελευθεροποίησης. Θα πρέπει να πιέσουμε στα θέματα αυτά και περιμένοντας το άνοιγμα αυτό θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας έτσι ώστε να, υπάρχει, να εφαρμοστεί και η αρχή της αμοιβαιότητα και θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες πρακτικές πλέον να δοθεί μια πρακτική και συνέχεια και να μην μένουμε μόνο στα θέματα αρχής. Θα πρέπει βεβαίως να ρυθμιστεί ένας ρυθμιστής ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο με ε, αρμοδιότητες και εξουσίες ε, πολύ πιο συγκεκριμένες από αυτές που αναφέρονται στο κείμενα που, έχουμε, που μελετάμε. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει και ένας ευρωπαϊκός οργανισμός για την έγκριση του υλικού που κυκλοφορεί. Ε, είναι και θέμα ασφάλειας ε, αλλά και είναι και θέμα ευθύνης των εταιριών. Επίσης με τον τρόπο αυτό δεν θα υπάρχουν ε, τεχνικά προβλήματα τα οποία θα αποτελούν εμπόδιο στην ολοκλήρωση της αγοράς. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η ιδέα της Κομισιόν για τα περιορισμένα διόδια που θα ισχύουν για τις κάποιες τεχνολογίες, διαιτιές κτλ. Τώρα, όσον αφορά το unbundling και ολοκληρώνω την παρέμβασή μου, θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με ιδιαίτερο ρεαλισμό και προσοχή. Μία πλήρης αποδέσμευση, κυρίως όσον αφορά και τον ε, διαχειριστή των υποδομών, μπορεί να ε, συνεισφέρει στην αύξηση του κόστους και των δαπανών. Πάντως, συζητώντας στην Επιτροπή τα θέματα αυτά, νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποια λύση. Ευχαριστώ. Η κυρία Τικάου για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Σαρακιάν για την έκδοσή της. Αυτή είναι η διατύπωση. Θα πρέπει να μπορέσει να μας βοηθήσει να έχουμε σε μια ενιαία ε, αγορά των σιδηροδρομικών μεταφορών και θα πρέπει να βελτιώσει και όλο το σύστημα των υποδομών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναπτύξει πολύ τα σιδηροδρομικά της δίκτυα, δεδομένου ότι έχουμε ε, μικρή επικράτεια αν θέλετε, αλλά πάρα πολύ πυκνό δίκτυο το οποίο μπορούμε να αναπτύξουμε. Όπως λοιπόν και με τα διευρωπαϊκά δίκτυα σε άλλους ε, τομείς ε, θα θέλαμε να προτείνουμε όλες οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να συνδεθούν μεταξύ τους με τρένα υψηλής ταχύτητα. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι δίδονται ε, λυπή κονδύλια για την συντήρηση των έργων υποδομής ήδη των υπαρχόντων. Γι' αυτό διαπιστώνεται ότι μειώθηκαν και οι επιβάτες που χρησιμοποιούν τα τρένα. Υπάρχουν όμως σχετικά κονδύλια τα οποία θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για τους σιδηροδρόμους. Είναι λοιπόν σημαντικό να γίνει μία μελέτη επιπτώσεων για να ξέρουμε ποια ήταν ε, τα αποτελέσματα του τι έγινε μέχρι τώρα. Εγώ είμαι υπέρ μίας ε, ε, νιές ευρωπαϊκής ρυθμιστικής αρχής και πιστεύω ότι δεν θα πρέπει η Επιτροπή να αναθέτει σε εξωτερικούς φορείς ε, συνέχεια κάποια κομμάτια που αφορούν τους σιδηροδρόμους. Η πρόσβαση επίσης στην αγορά θα πρέπει να γίνει με κριτήρια ε, διαφάνειας. Επίση, ο αριθμό των εργαζομένων στον τομέα και η ποιότητα της εργασίας του θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ευχαριστώ κύριο Σασάντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα κύρια θέματα που ήθελα να θίξω τα έξαν οι προηγούμενοι συνάδελφοι. Θα κάνω μια παρατήρηση λοιπόν για κάποια θέματα που δεν ανέφερε κανείς. Μίλησε προηγουμένως η Επιτροπή για μειωμένες τιμές για κάποιους που χρησιμοποιούν τους σιδηροδρόμους. Τι είδους μειώσεις, γιατί είδους μειώσεις μιλούμε. Ξέρουμε ότι έχουν ε, στη διάθεσή τους ε, αρκετό τροχαίο εξοπλισμό και υλικό οι αλλά δεν τον χρησιμοποιούν ίσως σωστά. Ίσως ένα ανταλλακτικό πολλές φορές ε, που λείπει να χρειάζεται πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ για να αντικατασταθεί. Και για να μπορέσουμε για να ανακαινήσουμε το τροχαίο μας εξοπλισμό, δεν χρειάζεται ίσως να δίδονται όλο και φτηνότερες τιμές. Ίσως θα μπορούσαν να έχουν οι σιδηρόδρομοι πρόσβαση σε κοινοτικά κονδύλια για να μπορέσουν να αντικαταστήσουν κάποιους από τους εξοπλισμούς τους και το τροχαίο τους κυρίως εξοπλισμό με σύγχρονο. εξοπλισμό. Ξέρουμε ότι οι διάφορες συμβάσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές στον τομέα αυτό για τον εξυγχρονισμό των σιδηροδρόμων. Αλλά το θεωρώ σημαντικό το θέμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε τελικά ο σιδηρόδρομος τι στόχο έχει, γιατί ασχολιόμαστε με αυτό το χώρο, για να βελτιώσουμε τις ε, υπηρεσίες που παρέχονται στους επιβάτες προφανώς σε ολόκληρη την Ευρώπη αυτό προσπαθούμε να κάνουμε από την άλλη μεριά όμως ξέρουμε ότι είναι τελείως κατακαιρματισμένες οι αγορές διαφορετικές οι δομές διαφορετικές οι υποδομές και από τεχνική άποψη ε, εδώ επιχειρείται μία με την αναδιατύπωση μία ενός είδους ενοποίηση η οποία όμως δεν μπορεί να γίνει πάση θυσία. Σε γενικές γραμμές, εκείνο που λέω ιδιαίτερα για το unbundling είναι ότι επί ουδελή λόγο θα μπορούσαμε να το δεχτούμε. Ε, ε, δεν είναι ε, το τίμημα που θέλουμε να πληρώσουμε για να φτιάξουμε ένα πιο ενιαίο, αν μάλλον πιο ενοποιημένο σιδηροδρομικό χώρο. Και ευχαριστώ την εισηγήτρια. Και εγώ ευχαριστώ. Η κυρία ντουρο απεσύρθη. Τελικά να πω εγώ μερικά λόγια να πω ότι στην συγγήτρια τη η δουλειά που έκανε είναι πάρα πολύ καλή και το βλέπουμε από α, τη συζήτηση που έγινε εδώ Το φαίνεται και από τη συζήτηση που γίνεται και εκτός ε, και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε έγγραφα σαν και τούτο εδώ που να πραγματεύουν τους σιδηρόδρομους και παρόλα αυτά να δημιουργούν ζωηρές συζητήσεις. Ή... Ακούστηκαν κάποια θέματα ε, προτεραιότητας. Εγώ είχα την εντύπωση ότι όλοι είχαμε συμφωνήσει για το unbundling, είχαμε ψηφίσει πρόσφατα υπέρ του unbundling. Οπότε με μπερδέψαν εκείνοι οι συνάδελφοι που λέει, πήραν το λόγο και είπανε «Ναι, όχι δεν θέλουμε το unbundling. Σας το υπενθυμίζω απλώς, κάντε ό,τι νομίζετε. Και κάτι άλλο, σε τελευταία ανάλυση κάποια στιγμή θα πρέπει η ενιαία αγορά, η εσωτερική αγορά να φτάσει και στο σιδηρόδρομο. Και εκείνο που με ανησυχεί είναι αυτό που είπε ο Ντέρκ Στέρκ. Να κάνουμε ορισμένα πράγματα. Μην έρθουμε μετά από δύο χρόνια και ζητούμε να γίνει πάλι αναδιατύπωση της αναδιατύπωσης και στην άλλη θητεία το ίδιο ξανά αναδιατύπωση. Και όταν είμαστε όλοι δυο μέτρα κάτω από το χώμα οι απογονοί μας θα έρθουν να κάνουν και αυτοί αναδιατυπώσεις και συνεχώς το Ευρωκοινοβούλιο να ζητάει, να ζητάει, να ζητάει αναδιατυπώσεις ή και πράγμα, αλλαγές και τα λοιπά και όταν βρίσκεται ενώπιον μια στρατής κατάσταση και αυτή στην οποία βρισκόμαστε σήμερα να σηκώνει τα χέρια ψηλά και να λέει θα δούμε Λοιπόν, σας ζητώ να επιδείξετε λίγο θάρρος, να διαβάσετε ακριβώς τι λέει η συγγήτρια στο εγγραφό της. Εγώ πραγματικά θέλω να δώσω τώρα το λόγο στην Κομισιόν για να ακούσω τι θα πει και η Κομισιόν, να ακούσω βεβαίως και την συγγήτρια και ε, πραγματικά πρέπει να σε πω και κάτι άλλο. Μας χρειάζεται διαφάνεια. Αυτή τη στιγμή η διαφάνεια δεν υπάρχει. Ο κύριος Πασκαρέλη πόσο, ένα λεπτάκι θέλετε, 30 δευτερόλεπτα. Αν μου δώσετε ένα λεπτό τότε να πω ότι η Κομισιόν επιβεβαιώνει την πρότασή της και επιμένει στην πρότασή της. Αν μου δώσετε παραπάνω χρόνο να απαντήσω και τις ερωτήσεις που γίνανε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, κυρία Σακαρέλια και όλους τους ομιλητές. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι για την πρόταση αναδιατύπωσης η Κομισιόν θέλει να εξασφαλίσει τη βέλτιστη λειτουργία του συνδρομικού δικτύου, βελτιώνοντας και όχι ε, αλλάζοντας ριζικά το όλο πλαίσιο ε, θα αφήσουμε την νομοθεσία ως έχει εκεί που δεν πρέπει να επαναδιατυπωθεί και ε, ούτω ή άλλω ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι 13 κράτη-μέλη βρίσκονται ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Η Κομισιό σε μια ανακοίνωσή της, ε, την οποία παρουσιάσαμε ταυτόχρονα με την πρόταση επαναδιατύπωσης, ότι θα αλλάξουν κάποια πράγματα αργότερα. Αυτό όχι γιατί θέλουμε κάθε δύο χρόνια να κάνουμε μια νέα αναδιατύπωση, αλλά είναι η φύση των πραγμάτων. Ε, η πραγματικότητα ε, τροποποιείται, εξελίσσεται, άρα και η νομοθεσία πρέπει να ακολουθεί. Το ίδιο γίνεται και με τις ε, συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε, κάθε τρία-τέσσερα χρόνια έχουμε και μια νέα συνθήκη. Το δεύτερο, η δεύτερη παρατήρηση που θέλω να κάνω είναι ότι η έκθεση Σερακιάνη στηρίζεται και το έχουμε πει πάρα πολύ στο ψήφισμα το οποίο θετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο πριν από μερικούς μήνες όπου ε, εκεί διαπιστώθηκε μια μεγάλη θα έλεγα σύμπτωση απόψεων με την Κομισιό και ε, η, η πρόταση για την επανατύπωση επαναλαμβάνει πολλά από τα θέματα τα οποία είχαμε θίξει και στο ψήφισμα. Επίσης, όσον αφορά για την πρότασή μας για τον ρυθμιστή, πρόταση για την οικονομική ρύθμιση των, της βιομηχανίας των δικτύων, ε, έχουμε ρυθμιστές που ήδη υπάρχουν, έχουν ε, αρμοδιότητες και εξουσίες πολύ διαφορετικές από στα κράτη-μέλη, στα διαφορετικές στα διάφορα κράτη-μέλη. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε σε όλους μεγαλύτερη ε, ανεξαρτησία και αποτελεσματικότητα και μεγαλύτερες αρμοδιότητες και επίσης να έχουν πρόσβαση και στις ε, συνδεδεμένες, στις συναφείς υπηρεσίες. Μιλάμε επίσης ε, σε μία, για μια θεσμοθέτηση του ρόλου του ρυθμιστή στην Ευρωπαϊκή Ένωση όντως ο συντονισμός, η ανταλλαγή απόψεων και ιδεών είναι κάτι που ευνοεί η Κομισιό με τον κανονισμό ε, που ήδη μόλις υιοθετήθηκε για τους διαδρόμους για τα εμπορεύματα ε, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι όντως χρειάζεται ένας ρυθμιστής ε, ε, για κάθε διάδρομο, αν θέλετε. Εγώ θα ήμουν ιδιαίτερα προσεκτικός στον παραλληλισμό που γίνεται ε, με τους τομείς που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει Ευρωπαίος ρυθμιστής. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε παραλληλισμούς ανάμεσα στην, ε, στις μεταφορές και στην ενέργεια. Για την ας πούμε, τηλεπιονής υπάρχει ένα σώμα, το body. Στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες υπάρχουν εθνικές υπηρεσίες. Άρα ένας Ευρωπαίος ρυθμιστής δεν μπορεί να αποφασίσει εκτός των διαδρόμων. Γι' αυτό προβλέπεται και από τον κανονισμό που μόλις συζητήθηκε. Κατά την άποψή μου, επομένω, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ε, στο ότι στο σιδηροδρομικό δίκτυο υπάρχει ε, φυσική ε, σύνδεση ανάμεσα στο τροχαίο υλικό, στο δίκτυο και στους ρυθμιστές. Ε, αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό των, ε, του συνδρομικού δικτύου. Θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε τα θέματα που αφορούν την πρόσβαση στην αγορά, την ανταγωνιστικότητα και με τα θέματα τα τεχνικά, δηλαδή η έγκριση ε, του τροχαίου υλικού λοιπά Αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Είναι θέμα οικονομικό και υπεύθυνο είναι, υπεύθυνες είναι οι εθνικές υπηρεσίες, ε, η, ασφάλεια και αυτό είχε δημιουργηθεί και από το τέταρτο συνδρομικό πακέτο το 2006-2007 και όλα αυτά συντονίζονται από την Ευρωπαϊκή Συνδρομική Υπηρεσία. Αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο θα επανέλθουμε το 2012 και είναι παράλληλα, παράλληλο με την ε, οικονομική και νομική ρύθμιση. Συναφές αλλά ξεχωριστό. Για την ε, τιμολόγηση, για, το, για την ε, δημοσιονομική ιεραρχία, αν θέλετε, του, στους Μιλάμε για τους διαχειριστές των υποδομών. Οι μεγάλες υποδομές ε, στα κράτη-μέλη ανήκουν ε, στα κράτη στα, ε, οι δημόσιες συγγνώμη, υποδομές, οι μεγάλες υποδομές ανήκουν στα κράτη-μέλη. Εξού και πρέπει να υπάρχει μια σαφής και σταθερή σχέση και σε σχέση ανάμεσα στους ε, μόνιμη σχεδόν σχέση ανάμεσα στον διαχειριστή και στις δημόσιες αρχές και πρέπει να υπάρχει μια απόλυτη διαφάνεια στις, ε, ε, στις χρηματοδοτήσεις έτσι ώστε να μην υπάρχει διπλή, να μην υπάρχει επικάλυψη. Είπαμε για τα μπόνους για στα RTMS και τα κίνητρα τα οποία ε, δίδονται για την επιλογή ε, βαγονιών που δεν ε, προκαλούν ιδιαίτερο θόρυβο, τα θόρυβα βαγόνια. Αυτό είναι θέμα που, με το οποίο ασχολείται η επαναδιατύπωση. Επίσης, προβλέπουμε και μια εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κόστους, θέμα το οποίο συζητήσατε και σήμερα το πρωί με την Ευρωβινιέτα. Είναι υπάρχει αυτή η σχέση ανάμεσα στα κείμενα. Επίσης θέλουμε να προωθήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο το Ευρωπαϊκό Σύστημα Σηματοδότησης, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ποιος πληρώνει όλα αυτά, όσες τις εκπτώσεις. Η λύση δεν επιβάλλεται από την Κομισιό. Η λύση μπορούμε να έχουμε ένα σύστημα μπόνους μάλους, όπως με τις ασφάλειες των αυτοκινήτων η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία θα αποφασίσει ή μπορεί να ε, αναλάβει την ευθύνη το κράτος που είναι και υπεύθυνο για την ε, οικονομική ισορροπία του διαχειριστή των ε, υποδομών. Δεν μιλάμε όμως για τεράστια ποσά τα οποία θα δαπανώνται, απλώς θέλουμε να δοθούν κάποια κίνητρα για να βελτιωθεί η κατάσταση. Μιλήσαμε για την δημοσιονομική αρχιτεκτονική που πρέπει να είναι στέρεη και που θα μας επιτρέπει να υπάρχουν φρέσκα κεφάλαια και να εξασφαλίσουμε και τις θέσεις απασχόλησης. Ε, σε, για να απαντήσω και στις, ε, παρεμβάσεις που ακούστηκαν ε, για την ε, απασχόληση στους σιδηροδρόμους. Βέβαια, ε, θα πρέπει να έχουμε και μια υποδομή στέρεα που να επιτρέπει να γίνονται επενδύσεις και θα πρέπει και ο σιδηρόδρομος να είναι ανταγωνιστικός σε σχέση με τις άλλες, άλλα μέσα μεταφοράς. Τώρα για τις συναφείς υπηρεσίες, τα rail-related services. Αυτό είναι ένα σημείο κλειδί των προτάσεών μας. Όπως σας είπα, θέλουμε να διευρύνουμε τις αρμοδιότητες του ρυθμιστή και στα θέματα των συναφών υπηρεσιών. Και θα ήθελα να τονίσω τέσσερις καινοτομίες τις οποίες εισάγουμε στην πρόταση. Καταρχάς την ανεξαρτησία του, ε, αυτού ο οποίος ε, έχει την ε, επιχείρηση, τη συνδρομική επιχείρηση αν θέλετε, σε σχέση με το δίκτυο, συνδρομικό δίκτυο. Στην νομοθεσία ο διαχειριστής των υποδομών είναι ανεξάρτητος σε σχέση με τις συνδρομικές υπηρεσίες. Όμως θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και την ανεξαρτησία του παρόχου των συνδρομικών υπηρεσιών. Γιατί αυτός ο πάροχος των συνδρομικών υπηρεσιών κάποιες φορές είναι και συνδρομική επιχείρηση ίδια. Ε, και αυτό θα πρέπει να το σπάσουμε γιατί εμείς λέμε ότι αυτός ο οποίος παρέχει τις συναφείς υπηρεσίες θα πρέπει να έχει τις ίδιες εγγυήσει ε, ανεξαρτησίας με αυτές που έχει ο διαχειριστής των υποδομών. Νομική ανεξαρτησία, ανεξαρτησία για τη λήψη αποφάσεων και οργανωτική ανεξαρτησία. Τώρα για τις ε, συναφείς υπηρεσίες επίσης το θέμα της αντιστροφής ε, του βάρους απόδειξης, ε, δηλαδή θα πρέπει αυτός να αποδείξει το, την ύπαρξη εναλλακτικών τρόπων και μέσων, όταν αρνείται δηλαδή την πρόσβαση στις συνδρομικές υποδομές. Εάν μία τώρα μία συνδρομική η υπηρεσία δεν χρησιμοποιείται για δύο χρόνια, ας πούμε, όπως λέμε στην πρότασή μας, τότε αυτός που το διαχειρεί, δεν μπορεί να το κλείσει. Πρέπει ή να το χρησιμοποιήσει ή να δεχτεί άλλοι, άλλοι ανταγωνιστές του μπορούν να το νοικιάσουν, να τον υπενικιάσουν και να το χρησιμοποιήσουν. Και αυτό για να μην κλείσει η αγορά. Επίσης, θα ήθελα να θίξω τώρα το πιο ευαίσθητο σε θέμα που είναι το unbundling που είναι η πλήρης αποδέσμευση ανάμεσα στην επιχείρηση, τη συνδρομική επιχείρηση και τον ρυθμιστή των συνδρομικών υπηρεσιών ε, και τον, ε, αυτόν που, ε, τον, τον ιδιοκτήτη, αν θέλετε, το, το δίκτυο, το συνδρομικό δίκτυο αυτό κάθε αυτό. είναι ακριβέ να πούμε ότι αυτή είναι η κατάσταση που ισχύει στην ενέργεια και στην, στις Δεν ισχύει. Για το συνδρομικό δίκτυο η Κομισιό έχει κάνει ε, άλλες επιλογές. Στο πρώτο πακέτο, το 2001, καταλήξαμε σε μια πολιτική συμβαστική ε, λύση, η οποία ήταν πολύ δύσκολη και πολύ ευαίσθητη. Εμείς είπαμε ότι δεχόμαστε αυτό το συμβιβασμό επί του παρόντος, θέλουμε όμως αυτό η συμβαστική πρόταση, η συμβαστική λύση να λειτουργήσει. Γι' αυτό ακριβώς ε, προσφύγαμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αντίον κάποιων κρατών μελών, διότι υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη που δεν σέβονται αυτό, αυτή τη συμβαστική πρόταση του 2001, όπου σύμφωνα με την λύση αυτή, ανεξάρτητα από το πώς λειτουργεί, ε, ποια είναι η επιχειρησιακή δομή του, της συνδρομικής εταιρείας ε, ή των, ε, των σιδηροδρόμων, θα πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός. Εκεί που υπάρχει holding, στις χώρες που υπάρχει holding, holding δεν, 6 ε, σε 7 περιπτώσεις δεν υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο κατα, ε, καταφύγαμε, προσφύγαμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι λέει το δικαστήριο ή τι θα πει το δικαστήριο πάνω σε αυτό το σημείο και είμαστε όμως βέβαια και ανοιχτοί ταυτόχρονα να δούμε τι θα αποφασίσει και ο νομοθέτης. Νομοθέτης που είναι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Επίσης, όσον αφορά... Ε, ήθελα να πω ότι η σιδηρόδρομη είναι πάρα πολύ περίπλοκο θέμα, όχι μονάχα για τις αποφάσεις στις πολιτικές που πρέπει να ληφθούν, αλλά και για τεχνικές αποφάσεις. τεχνικές αποφάσεις που, πρέπει να, που στηρίζονται στις πολιτικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί πιο πριν και που πρέπει να ληφθούν και πάρα πολύ γρήγορα. Πρέπει να δούμε τι, λαμβάνοντα υπόψη αυτό που επιτρέπει η συνθήκη της Λισαβόνας, είπαμε να ε, έχουμε την δυνατότητα μέσω ε, πράξεων, αν θέλετε, ε, κάποιων πράξεων, να τροποποιήσουμε τα παραρτήματα. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να υπαναχωρήσουμε στο σημείο αυτό, διότι αλλιώς θα έχουμε την ε, διαδικασία συναπόφασης, ενώ αυτού του είδους παρακτήματα μπορούν να τροποποιηθούν ε, με έναν ε, απλό τρόπο, με την επιτροπολογία, ας πούμε, που είναι πιο σύνηθες. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος ο πρόεδρος. Η κυρία Σερακιάνη θα ήθελε να προσθέσει κάτι. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Πρόεδρε, σπάνια νομίζω ότι έχω προκαλέσει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον και θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν στην συζήτηση για το ενδιαφέρον που έδειξαν γιατί πιστεύω ότι από αυτή την πολύτιμη ε, συνεισφορά τους θα γίνουν οι καλύτερες επιλογές ε, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε, τα, ή όμως νομίζω θα έπρεπε να υπογραμμίσουμε τα βασικά στοιχεία του working document. θα ήθελα να κάνω όμως μερικές παρατήσεις, πολιτικού χαρακτήρα ενδεχόμενα, αλλά τέλος πάντων παρατηρήσεις τις οποίες θα πρέπει να έχουμε κατά νου σε αυτή τη συζήτηση που κάνουμε. Τρεις, τρία στοιχεία που πρέπει να τα σκεφτούμε. Το ένα είναι ότι όντως οι μεταφορές εμπορευμάτων αποτελούν μια αγορά που ο σιδηρόδρομος είναι στο 11% ενώ οι επιβάτες είναι 6%. Επομένως ο σιδηρόδρομος έχει προβλήματα, αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα θα έλεγα και κάποια κράτη θα πρέπει να ε, παρέμβουν, να, εφαρμόσουν, να προχωρήσουν σε κάποιες χρηματοδοτήσεις. Όπως είπε και η Κομισιόν, 13 είναι οι παρεμβάσεις ε, που έγιναν ε, σε σχέση, σε σχέση με το, πρώτο, με το προηγούμενο πακέτο και έχουμε 25 μοντέλα σιδηροδρομικών ε, δικτύων. 25 έχουμε γιατί η Μάλτα και η Κύπρος δεν έχουν σιδηροδρόμους, αλλιώς είχαμε 27. Λοιπόν, Αυτά τα τρία στοιχεία θα πρέπει να τα έχετε κατά νου για να, και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να είμαστε φιλόδοξοι. Καλό είναι να είμαστε και συνετοί και προσεκτικοί κτλ. Όμως εγώ σας καλώ να είμαστε φιλόδοξοι γιατί ο καθήκον μας είναι να βρούμε μια λύση σε ένα σύστημα το οποίο αντιμετωπίζει δυσκολίες. Προφανώς αυτές είναι μόνο προτάσεις και ε, πραγματικά καλωσορίζω τις προτάσεις που έκαναν οι συνάδελφοι και η Κομισιόν και εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να το διευρύνουμε αλλά όλα αυτά και στο εθνικό επίπεδο ε, και θυμάμαι και ότι υπήρχαν κάποια κίνητρα τα οποία, κάποιες προτάσεις που έγιναν για να, και για τον Ευρωπαίο ρυθμιστή ε, και ιδίω στην πρώτη φάση είχαμε πει να υπάρξει ένας εθνικός ρυθμιστής που να έχει την, τους απαραίτητους ανθρώπινους οικονομικούς πόρους, ανεξαρτησία κτλ. και να δημιουργηθεί ένα δίκτυο ρυθμιστών αλλά και γιατί να μην έχουμε και τον Ευρωπαίο ρυθμιστή Επίση να πω ότι η συζήτηση για τον Ευρωπαίο Ρυθμιστή είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι αν δεν καταφέρουμε να έχουμε μια ισχυρή φιγούρα, ε, μια ανεξάρτητη φιγούρα, τότε δεν μπορούμε να συζητήσουμε το unbundling, διότι αν έχουμε το πρώτο κομμάτι, αν θέλετε, της επαναδιατύπωση. θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να εφαρμόσουμε και όλα τα τριγύρω, τα οποία ε, αποτελούν και τη βάση για την πρόταση τη Κομισιόν. Για τη χρηματοδότηση, προφανώ ε, όλοι συμφωνούμε ότι αυτό το σύστημα πρέπει να εφαρμοστεί και επαναλαμβάνουμε επαναλαμβάνω ότι η πρόταση ε, των πενταετών προγραμμάτων ε, σχεδίων θα πρέπει να τύχει υποστήριξη και όλοι συμφωνούν ε, για τα θέματα ασφάλειας και επιστοποίησης. Και αυτό δεν έχει να κάνει με την επαναδιατύπωση. Αν θέλουμε όμως να είμαστε φιλόδοξοι, μπορούμε να έχουμε και, κάποιες, ε, και κάποια θέματα στην επαναδιατύπωση για να δούμε τι θα γίνει το 2012. Δηλαδή αν κάνουμε καλά τη δουλειά μας τώρα θα μπορέσουμε να είμαστε πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι όταν έρθει η ώρα να κάνουμε την ελευθεροποίηση, την, να στήσουμε θέματα ασφάλειας κτλ. Λυπάμαι που ο κύριος Στέρξ έφυγε, και, αλλά το λέω και στην Κομισιό. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν, ε, ότι περιμένουμε ε, τις αποφάσεις του δικαστηρίου. Όμως πιστεύω ότι στις επιλογές που πρέπει να γίνουν, πρώτο, καθεδρία έχουν, ε, έχει πολιτική αν θέλετε. Ε, επομένως δεν θα πρέπει να περιμένουμε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Δεν είναι οι δικαστέ που θα επιβάλλουν τους κανόνες σε μια ενιαία αγορά που εμείς θα πρέπει να ε, καθορίσουμε και τα σημεία, τα βασικά σημεία τη θα πρέπει εμείς να, να καθορίσουμε. Γι' αυτό θα πρέπει να ε, προωθήσουμε ένα φιλόδοξο σχέδιο ε, το οποίο αναφερόταν και στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το, του Ιουνίου του 2010, όπου θίγαμε διάφορα σημαντικά θέματα, συγκεκριμένα και αυτή την, το διαχωρισμό, την αποδέσμευση. Εγώ θέλω να είμαστε ε, ρεαλιστές. Ε, για, αυτή την, ε, για την αποδέσμευση, εγώ δεν θα έδινε και τη ζωή μου. Όμως θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, διότι πιστεύω ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες συνθήκες, έτσι ώστε να μην επιλέξουμε απλώς ένα από τα συστήματα, από τα 25 ε, τα οποία είναι διαθέσιμα, δηλαδή να διαλέξουμε το γερμανικό μοντέλο σε εις βάρος του Ιταλικού ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Όχι, θα πρέπει να επιλέξουμε τα καλύτερα στοιχεία, τις βέλτιστες πρακτικές και αυτές οι βέλτιστες πρακτικές θα πρέπει να ε, εφαρμοστούν ε, σε όλα τα κράτη-μέλη. Ένας από αυτούς τους κανόνες πρέπει να είναι και η αποδέσμευση, ε, ο διαχωρισμός. Πρέπει να δούμε όμως τι ακριβώς είδους αποδέσμευση ή διαχωρισμό χρειαζόμαστε. Πιστεύω ότι μια τέτοιου είδους επιλογή που ε, είναι πάρα πολύ σημαντική, πρέπει να την, την απόφαση για αυτή, την, για αυτή, για αυτή την, ε, αυτό το διαχωρισμό πρέπει να, τον πάρει, να την πάρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και ολοκληρώνω, πρόεδρε, να πω ότι εγώ μπορεί να είμαι νέα πρόεδρε, αλλά δεν θέλω μετά από 10 χρόνια να είμαι εδώ και να συζητάμε την επαναδιατύπωση της, αναδιατή, της επαναδιατύπωσης. Γι' αυτό θα ήθελα να βρούμε ε, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε όσο να δω καλύτερα το σιδηρονομικό δίκτυο. Δεν λέω να κάνουμε μια επανάσταση. Εγώ λέω να βελτιώσουμε το θέμα και δεν θα πρέπει να χάσουμε την ευκαιρία που μας προσφέρετε τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Σέρα και Είσαστε οι νεότεροι μεταξύ ημών. Επομένως θέλουμε κατά τη διάρκεια της δικής σας ζωής τουλάχιστον να γίνουν όλα αυτά. Να υπενθυμίσω στα μέλη ότι το σχέδιο έκθεσης θα το έχουμε στη διάθεσή μας τον Μάρτιο. Τον Μάιο θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή Μεταφοράς και θα περάσει από την Ολομέλεια του Ιουλίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το έγγραφο εργασίας και για την συζήτηση. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Ωραία, τελειώσαμε συνάδελφοι για σήμερα στις 9 η ώρα. Έχουμε διάφορα θέματα που θα μας ε, απασχολήσουν. Θα τα πούμε αύριο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και όλους τους γερμηνείς. Ε, καλό σας βράδυ.